Ας ξεκινήσουμε, παρακαλώ πολύ. Καθίστε. Και οι Πολωνοί εκπρόσωποι επίσης, οι εκπρόσωποι της Πολωνικής Αντιπροσωπείας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε σήμερα την, επίσης, το επίσημο ξεκίνημα της Ιρλανδικής Προεδρίας στην Επιτροπή μας. Είμαστε σε επαφή από τις αρχές Ιανουαρίου με την Ιρλανδική Προεδρία, αλλά για πρώτη φορά σήμερα έχουμε τον Υπουργό Μπρένταν Χάουλιν, Προεδρεύων του Συμβουλίου, υπεύθυνο για την πολιτική συνοχή. Ο κύριος Χάουλιν είναι Υπουργό Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρύθμισης. Θέλετε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να απευθυνθώ και στον κύριο Βανίστε Ρόι και πραγματικά να πω ότι η γραβάτα η οποία φοράει είναι πραγματικό δείγμα αλληλεγγύης προς την ε, Ιρλανδική Προεδρία, καθότι είναι η γραβάτα της Ιρλανδικής Προεδρίας. Προσβλέπω σήμερα σε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε έναν τομέα της δημόσιας πολιτικής που πραγματικά πιστεύουμε όλοι ότι βρίσκεται στην καρδιά της επιστροφής της Ευρώπης στην οικονομική ανάκαμψη. Τους τελευταίους μήνες, προετοιμάζοντας την Προεδρία της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο των Υπουργών, είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ μαζί σας, κυρία Πρόεδρε, αλλά να συναντήσω επίσης και πολλούς εισηγητές υπεύθυνου για το νομοθετικό πακέτο της συνοχής. Θεωρώ ότι οι συζητήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές και πραγματικά θα ήθελα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία τη επίσκεψή μου στι Βρυξέλλε αυτή την εβδομάδα για να συνεχιστεί αυτό ο διάλογο, αυτή η συνεργασία που θεωρώ ότι πραγματικά είναι ιδιαίτερα αξιόλογη, καθότι πραγματικά μα βοηθά και του μεν και του δε να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά πώ πρέπει να συνεργαστούμε κατά τη διάρκεια τη Ιρλανδική Προεδρία. Προσβλέπω λοιπόν σε μια στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου και εσά, μέλη τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη του Κοινοβουλίου, του επόμενου έξι μήνε. Το 2013 είναι η 40η επέτειος της προσχώρησης Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, όπως ονομαζόταν τότε. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να αναπτυχθεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά η Ιρλανδία στις δεκαετίες που μεσολάβησαν. Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε πραγματικά ένα πολύ βασικό εταίρο στο πρόγραμμα ανάκαμψης Ιρλανδίας αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη πρόκληση προσπαθώντας να βελτιώσουμε την οικονομία μας και τα δημόσια οικονομικά μας. Προκειμένου όμως να ανταποκριθούμε στην... Μάλλον θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή και είμαι σίγουρο ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε την Ιρλανδία πίσω σε μια κατάσταση θετικής οικονομική ανάπτυξη με μεγάλη απασχόληση. Θεωρεί η κυβέρνηση τη Ιρλανδία ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ζωτική για την οικονομική μας ανάκαμψη και το μέλλον της χώρας μας. Παραμένουμε ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε το κοινοτικό έργο. Πολλά έχουν αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που προσχώρησε η Ιρλανδία το 1973. Όχι μόνο διευρύνθηκε από 9 σε 27 κράτη-μέλη, σύντομα 28, αλλά η ίδια η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διευρυνθεί και έχει εμβαθυθεί μία από τις βασικές εξελίξεις ήταν ε, ο δυναμωμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός ο δυναμωμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά χαιρετίζω ιδιαιτέρως. Μιλάω σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ως βουλευτής και ο ίδιος. Τον επόμενο μήνα κλείνω 30 χρόνια περίπου στο Ερλανδικό Κοινοβούλιο και μάλιστα υπήρξα βουλευτή τόσο στην κάτω όσο και στην πάνω βουλή και μάλιστα υπήρξα και αντιπρόεδρος τη κάτω βουλής της ΔΑΕΛ. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική και ουσιαστικά την χρησιμοποιώ και την εκμεταλλεύομαι στο νέο ρόλο που έχω ω Υπουργό Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρύθμιση. Πρόκειται για ένα νέο Υπουργείο που προβλέπεται στην Ιρλανδική κυβέρνηση. Στα πλαίσια λοιπόν των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμόσω, θα ήθελα να εξυγχρονίσω τη λειτουργία του Εθνικού μα Κοινοβουλίου, ιδίω όσον αφορά τι κοινοβουλευτικέ εξεταστικέ επιτροπέ, προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και να βαθμίσουμε το ρόλο των βουλευτών. Μετά την οικονομική αυτή κρίση, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν για τα συστήματα διακυβέρνηση και πιστεύουν ότι αυτά θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Στο ίδιο πνεύμα, δίνω ιδιαίτερη αξία σε όλε τι αλλαγέ που έχουν γίνει προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στο νομοθετικό πλαίσιο για πάρα πολλέ πολιτικέ όπω η πολιτική συνοχή. Ο ρόλο αυτό φέρνει πραγματικά την Ευρώπη πιο κοντά στου πολίτε τη, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε, ιδίω το 2013 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτο του Πολίτη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κατά την προετοιμασία τη Ιρλανδική Προεδρία το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα να συναντήσει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, και επίση η κυβέρνησή μας είχε τη δυνατότητα να συναντήσει τη διάσκεψη των πρόεδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ο ίδιος θα παραστώ σε αυτή τη διάσκεψη πολύ σύντομα. Πραγματικά, οι συναντήσεις αυτές δημιούργησαν ένα πολύ θετικό πνεύμα συνεργασίας. Και στη ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου θα συνεχίσουμε τη στενή αυτή σχέση. Το 2013 επίσης σηματοδοτεί την 7η φορά που η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευκαιρία την οποία θέλει να εκμεταλλευτεί η Ιρλανδική κυβέρνηση αλλά και οι άνθρωποι της Ιρλανδίας. Η Προεδρία Τη Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά αποδεικνύει τελικά ότι μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση που περιλαμβάνει μεγάλε και μικρέ χώρε. Το γεγονό ότι μια μικρή χώρα σαν την Ιρλανδία μπορεί να δραματίσει ένα πολύ σημαντικό κεντρικό ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι κάτι πολύ σημαντικό που πραγματικά τονίζει τη διαδικασία εμβάθυνση και διεύρυνσης Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολονότι είχαμε επιτυχίε στο παρελθόν, θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή βασίζεται μόνο σε σκληρή δουλειά και σε δέσμευση. Η Προεδρία δίνει τη δυνατότητα στην Ιρλανδία να αποδείξει ότι αποτελεί ένα αφοσιωμένο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά ανήκει στην καρδιά λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία ανακάμπτει και η οποία θα βοηθήσει την οικονομική ανάκαμψη τη Ευρώπη. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία με του εταίρου μα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει από την κρίση αυτή ακόμα πιο δυνατή αλλά δεν υπεκτιμούμε σε καμία περίπτωση την πολύ σκληρή εργασία την οποία πρέπει να επιτελέσουμε. Θέλουμε η Προεδρία μας να είναι πραγματικά δίκαιη, ειλικρινής, λειτουργική και θα πρέπει πραγματικά να στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλουμε στενά να συνεργαστούμε με όλους μας τους εταίρους και με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε την ατζέντα μας επικοδομητικά και μέσω συνένεση. Η προσέγγιση αυτή ήταν ιδιαίτερα θετική τόσο για την Ιρλανδία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν και θέλουμε να τη συνεχίσουμε και κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2013. Στι επαφέ μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να εκφράσουμε κάθε φορά την πεσυμφωνημένη ε, θέση του Συμβουλίου με έναν τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση όμως τι εξουσίες Ευρωπαϊκή Ένωση ω νομοθέτη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συγχωρείτε ως νομοθέτη. Θέλουμε λοιπόν μια στενή και επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στι φιλοδοξίε μα. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την Προεδρία σε μια στιγμή πολύ μεγάλων προκλήσεων για την Ιρλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δραματίσει έναν ζωτικό ρόλο στη διαδικασία τη οικονομική ανάκαμψη όλων των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε κράτο μέλο ξεχωριστά. Η βασική στρατηγική προτεραιότητα για την Προεδρία μας είναι να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αύξησης ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Θέμα της Προεδρίας μας είναι η σταθερότητα, οι θέσεις εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας αναφέρεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις τις οποίες πρέπει να λάβουμε για να πετύχουμε τις βασικές προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας θα προευρεύσουμε και τις νέα διαφορετικές συνθέσεις του Συμβουλίου τους επόμενους έξι μήνες και θα έχουμε στενές συζητήσεις με το Κοινοβούλιο για όλα τα θέματα. Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές. Μία ανάκαμψη που να βασίζεται στους ανθρώπους και η οποία να είναι βιώσιμη. Επενδύσεις πρέπει να γίνουν σε ε, θέσεις εργασίας και στους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια γενικότερη δέσμευση με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Η χρηματοδότηση της συνοχής, όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά, στο κέντρο της ατζέντα μας για την οικονομική ανάπτυξη και πραγματικά θέλουμε να προωθήσουμε τις απενδύσεις που θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας στο μέλλον, προσπαθώντας να πετύχουμε παράλληλα τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια ευφυή βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Τα 40 χρόνια συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά καταδεικνύουν ότι η πολιτική συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς επίσης και της συνοχής. Και θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση, η συνοχή, οι δύο αυτές λέξεις έχουν ένα πραγματικό νόημα και πραγματικά έχουν συμβάλει στο να μειωθούν οι κοινωνικέ και οικονομικές αποκλήσει και στο να αυξηθεί ουσιαστικά και ειλικρινά η συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ένωση 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε 27 κράτη-μέλη σε 271 διαφορετικές περιφέρειες. Οι επενδύσεις που γίνονται από τον κοινοτικό προπολογισμό είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τα κράτη-μέλη και για τις μονομένες περιφέρειες και πραγματικά μπορεί να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη. Η εμπειρία της Ιρλανδίας στα πλαίσια τη συνοχή ήταν πάρα πολύ θετική. Η πολιτική συνοχή διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιρλανδικής οικονομία. Μπορούμε να πούμε ότι ένα καταπληκτικό παράδειγμα της πολιτικής συνοχής είναι το πρόγραμμα PIS. Ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά συνέβαλε πάρα πολύ στην μεθόριο της Ιρλανδίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στην ειρήνευση και τη συμφιλίωση στην Βόρειο Ιρλανδία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και στόχο του είναι να οδηγηθούμε σε μια ειρηνική και σταθερή κοινωνία και να προωθήσουμε τη συμφιλίωση μέσω δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν τη συμφιλίωση των κοινοτήτων και την ανταλλαγή εμπειριών για την κοινωνία και στις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν υπήρξε ένας πολύ ισχυρό υποστηρικτής τη Ειρηνή σε κάθε τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης όπως άλλωστε φαίνεται και από το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο αποδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι. Η νέα πολιτική συνοχή είναι πάρα πολύ στενά στεδεμένη με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα μία συμφωνία, συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σαφώ επηρεάζει την επεξεργασία του νομοθετικού πακέτου. Η Προεδρία προφανώς θα τηρήσει την συνήθη διαδικασία νομοθεσίας. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να πετύχουμε μια συμφωνία για όλο το νομοθετικό αυτό πακέτο κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας, δηλαδή τους επόμενους έξι μήνες. Και θεωρώ ότι και η δική σας Επιτροπή την ίδια φιλοδοξία έχει. Αυτό κατάλαβα από τις συζητήσεις που κάναμε. Η αξία του στόχου αυτού είναι πραγματικά ξεκάθαρη. Εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να δώσουμε στα προγράμματα αυτά την απαραίτητη νομική ασφάλεια προκειμένου τα προγράμματα της συνεχής να μπορέσουν να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά το 2014. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο έχει κάποιες γενικές εν μέρη προσεγγίσεις για κάποια θεματικά ζητήματα τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2012. Υπάρχουν ακόμα όμως κάποια ζητήματα τα οποία εκκρεμούν στο Συμβούλιο που έχουν να κάνουν με τις τελικές διατάξεις καθώς επίσης και την ευρωπαϊκή ομαδοποίηση της ε, εδαφικής ε, συνεργασίας και τον σχετικό τροποποιητικό κανονισμό. Ελπίζουμε ότι για τα εκκρεμή αυτά ζητήματα θα ληφθεί απόφαση στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Θα ήθελα επίσης ε, να τιμήσω ιδιαίτερα τη συνεισφορά της Δανικής και Κυπριωτικής Προεδρίας για τα επιτεύγματά του, για το ότι κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το πολύπλοκο αυτό νομοθετικό πακέτο. Θα ήθελα επίση να πω όμω ότι συνέβαλε πάρα πολύ και η Πολωνική Προεδρία, προσπαθώντα να πλαισιώσει νομοθετικά όλα αυτά τα ζητήματα ήδη από το 2011. Επίση, θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έγινε στο νομοθετικό, στην νομοθετική δέσμη μέτρων στο Κοινοβούλιο όπου η Επιτροπή Περιφερική ανάπτυξη κατέδειξε σε σχέση με το εύρο των νομοθετικών αυτών θεμάτων που εξαρτώνται από το ε, MFF ε, έχουν σημειώσει πρόοδο. Επιπλέον ένα σημαντικό μέρο τη πρόοδου έγινε στου τριμερεί διαλόγου που ξεκίνησαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Κυρίω όσον αφορά τον συμβιβασμό πριν από τα Χριστούγεννα για το στατηγικό πρόγραμμα των στοιχείων για τι κοινέ διατάξει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή τη διαδικασία φέτο βρισκόμαστε σε καλή θέση. Ωστόσο δεν θα ήθελα να υποβαθμίσω με κανένα τρόπο το τεράστι, τις τεράστιες προκλήσεις του έργου που αντιμετωπίζουμε αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες επί ενός νομοθετικού ε, πακέτου μέτρων ώστε οι εταιρικές συμφωνίες να μπορέσουν για τα λειτουργικά προγράμματα να είναι έτοιμες και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε, σε σχέση με τα 27 κράτη-μέλη, 28 όταν θα έρθει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό πανευρωπαϊκά για την πολιτική συνοχή και έχει τεράστια σημασία για τους πολίτες της Ευρώπης. Σημεριζόμαστε την ευθύνη και τον κοινό στόχο ως φιλοδοξία να καταλήξουμε σε συμφωνία το δυνατόν γοργότερα στο Συμβούλιο. Εμείς από πλευρά Συμβουλίου εκτιμούμε την ε, οικοδομητική, επικοδομητική προσέγγιση από το Ευρωκοινοβούλιο που ε, οδήγησε σε ένα συμβιβασμό όσον αφορά το στρατηγικό προγραμματισμό. Και οι δύο νομοθέτε, συνομοθέτε, πρέπει να συνεχίσουν αυτή την επικοδομητική συνεργασία. Από κοινού λοιπόν θα συνεργαστούμε ω συνομοθέτε με το Ευρωκοινοβούλιο για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι σε τριμερείς ε, διαλόγους με την Επιτροπή και με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με την Κυπριακή προεδρία έτσι θα συνεχίσουμε. Όπως και σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών αλλά πρέπει να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες σε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το καλοκαίρι. Η προεδρία, εγώ ο ίδιος, η, η δική μου υπάλληλη είναι στη διάθεσή σας πάντα και προσβλέπω στο να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική σας επιτροπή και να αναφέρω την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί υπό την Ιρλανδική Προεδρία. Εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία να προσφωνήσω την Επιτροπή σας. Λέμε στα Ιρλανδικά ως παροιμία Δύο άνθρωποι μπορούν να δουν και να κάνουν πράγματα τα οποία ένα δεν μπορεί. Υπό αυτό το πνεύμα λοιπόν προσβλέπω σε μια ανταλλαγή απόψεων επικοδομητική μαζί σας. Σα ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ Υπουργέ και όπως ήθιστε θα δώσω καταρχάς το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ο Λάμπερτ που φοράει και μια καταπληκτική γραβάτα ε, είναι, δεν έχει άλλη πλέον να ξεκινήσει. To, to have the speech of, of, the minister second to go after the, the, speech of Cameron this morning. So you didn't, Πρέπει να πω ότι ήσασταν πάρα πολύ συγκεκριμένος, θετικός, δεν είναι και εύκολο γιατί έπρεπε να πετάξει και να περάσει πάνω από τη θάλασσα για να έρθει στην Ευρώπη. Λοιπόν, πράγματι, ε, ακούσαμε πολύ καλά πράγματα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνεκτικότητα πιο πολύ. Αυτό μας απασχολεί και στην Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Και το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει και ένας επαρκής προϋπολογισμός, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι συμβεί θα είναι πολύ πιο πάνω από τα 300 εκατομμύρια ή μεγαλύτερα ποσά που θα διατεθούν για τα ταμεία μας. Και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ιδίω αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Και συγκεκριμένα τα μέσα τα οποία πλέον έχουμε στις νομοθεσίες. και δεν είναι ρόλος μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και της Κομισιόν και του Συμβουλίου όχι μόνο να πείσουμε αλλά και να κάνουμε τις χώρες να επιταχύνουν και την εκτέλεση των συμφωνιών εταιρική σχέσης. Το 2014, τους πρώτους μήνες, το πρώτο εξάμεινο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να είναι χαμένος χρόνος. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και να επιταχύνουμε. Και έτσι πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση. Στρέφομαι λίγο στο πρόγραμμά σας και κάτι λείπει, κάτι λείπει. Υπουργικές συναντήσεις είναι κρυμμένο κάπου στις γενικέ υποθέσεις. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω κάπου να συνεδριάζει το σώμα αυτό. Ξέρετε ότι έχουμε το πολιτές μουσιονομικό πλαίσιο και στο διαπραγματευτικό κουτί υπάρχουν ζητήματα που μας ενδιαφέρουν και αποτελούν και επίκεντρο των δικών μας εργασιών και του ρόλου, του ρόλου μας ως συνομοθετών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε και τι περιθώρια ελιγμών έχει το Συμβούλιο. Όταν θα έχουμε ένα πολιτές μεσονομικό πλαίσιο, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη διάφορα άρθρα. Για παράδειγμα, μακροαιρεσιμότητα, το μαθηματικό επίδοση, ε, θέματα όπως είναι η επιβολή των ορίων, το κάπινγκ και ούτω καθεξής υπάρχουν περιθώρια λιγμών και διαπραγματεύσεων. Διότι καλό είναι ο σεβασμό, αλλά αν υπάρχουν πιέσει ε, και ο χρόνο δεν περισσεύει, τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι να δούμε όλα αυτά τα σημεία κατά πόσον αν θέλει το Συμβούλιο να περιληφθούν στο πολιτισμικό πλαίσιο, μπορεί να αλλάξει αυτό. Εγώ θα ήμουν αντίθετο. Να δούμε λοιπόν τι περιθώρια έχουμε Γιατί και εμείς πρέπει να ολοκληρώσουμε για τη δουλειά που κάνουμε με την εξέταση των διαφόρων κανονισμών. Ίσως αυτή θα είναι τελευταία παρατήρηση, φαντάζομαι θέλουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Τι συνέργειες υπάρχουν μεταξύ των ταμείων. Η κυρία Γέγγεν Κουίν εργάζεται και αυτή για την ένωση της καινοτομίας την ανάπτυξη της έρευνας των συνεργειών και ούτω καθεξής. Στρέφουμε πάλι προς τη συζήτηση για το πολιτεύσιμο οικονομικό πλαίσιο. Αν δει κανείς τι γίνεται με το προπολογισμό για την έρευνα και την ανάπτυξη. Και συγκεκριμένα αν δούμε τις θεματικές προτεραιότητες μέσα από τα περιφερειακά ταμεία. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα για συνέργειες, σημαντικές συνέργειες στο τομέα της γνώσης, της έρευνας, των υποδομών έρευνας, της εκπαίδευσης, ιδίως από το Περιφερειακό Ταμείο. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό για να ε, είμαστε ανταγωνιστικοί και ισχυροί. Ιδίως έχοντας υπόψη ε, τη νέα γενιά που δυστυχώς ακόμη είναι εκτός αγοράς εργασίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα σχολιάσετε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως που ήρθατε εδώ. Και ναι πράγματι, όπως και εσείς και εγώ, είμαι πεπισμένος ότι στο εξάμεινο της Ιρλανδικής Προεδρίας θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Δεν μπορούμε, παραλαμβάνω, το 2014, πριν τις εκλογές, να πάμε στους πολίτες μας και να πούμε «Χάσαμε μια χρονιά» και δεν έχουμε μια πραγματική πολιτική συνοχή στου κανονισμού που να λειτουργεί, που να φέρνει αποτελέσματα. Όχι, δεν μπορούμε, δεν μπορώ να πάω να πω τέτοια πράγματα στους ψηφοφόρους μας. Τι ακούμε τι τελευταίε ημέρε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 7 και 8 Φεβρουαρίου πρώτα απ' όλα θα λάβει χώρα. Αυτό μας δίνει και κάποια ελπίδα ότι ίσω υπάρξει και εξέλιξη με το θέμα του πολιτού πλαισίου και αυτό αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για τις πολιτικές μας. Διότι δεν υπάρχει πολιτική συνοχής ε, χρόνο με το χρόνο. Δεν μπορούμε να τα αποφασίζουμε την τελευταία στιγμή. Σίγουρα χρειάζονται χρήματα, αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα είναι να έχουμε το σύστημα και να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθεί, να ληφθούν ε, έγκαιρα οι αποφάσεις και είμαι πεπισμένος ότι θα το πετύχουμε. Ναι, ας προχωρήσουμε, ας το κάνουμε λοιπόν. Thank you for all those commitments. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δεσμεύσεις που αναλάβατε, Λάμπερτ. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ουσιαστικά δεσμευτήκατε εσείς ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και επειδή θα προεδρεύω το τριμνούς διαλόγου θα σας πιέσω. <laughs> so now we need... Ελπίζω να γίνουν πράξη οι καλές ειδήσει. Για να πούμε, οι σοσιαλιστές θα πούν τα ίδια, ο Γιώργος Σταυρακάκης. Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ τόσο εκ μέρους της συντονίστριας της πολιτικής μου ομάδας, Κωνσταντζε Κρέλ, που δυστυχώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί στη σημερινή μας συνεδρίαση, όσο και από τη μεριά μου και εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, να καλωσορίσω την Ισλανδική Προεδρία του Συμβουλίου και εσάς προσωπικά στην Επιτροπή μας. Αναγνωρίζουμε ότι η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια κρίσιμη καμπή στι διαπραγματεύσει για το νομοθετικό πακέτο τη πολιτική συνοχή για μετά το 2013. Κατά τη διάρκεια του τριλόγου τη 19η Δεκεμβρίου, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ήρθαν σε συμφωνία για τον μπλοκ που σχετίζεται με το στρατηγικό σχεδιασμό που παρέχει στα κράτη-μέλη τη βεβαιότητα για την προετοιμασία των προγραμμάτων του. Με αυτόν τον τρόπο οι φορεί σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση μπορούν άμεσα και χωρί καθυστερήσει να ξεκινήσουν την προετοιμασία του για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το πνεύμα τη στενής επικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία ευελπιστούμε να συνεχιστεί έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει μέχρι το καλοκαίρι και η νέα πολιτική συνοχή να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ιρλανδική Προεδρία. Όπω αναφέρατε κι εσεί κύριε Υπουργέ, οι βασικέ αρχέ που διέπουν την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου είναι η σταθερότητα, απασχόληση και η ανάπτυξη. Και οι τρει αυτέ αρχέ απατώνται στην πολιτική συνοχή ω μια πανευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική η πολιτική συνοχή αποτελεί το κύριο επενδυτικό εργαλείο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την επίτευξη σταθερότητα μεταξύ των περιφερειών, την ανάκαμψη, την τόνωση τη ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία τέσσερων απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προτού ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, θα μου επιτρέψετε να σα θέσω ένα θέμα που μα απασχολεί από την αρχή των διαπραγματεύσεων για του κανονισμού και έχει να κάνει με το MFF. Γνωρίζουμε ότι ασχολείται ο κ. Βαν Ρομπάη, αλλά σαν Προεδρία έχετε το δικό σα ρόλο να παίξετε. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο για το Πολιετέ Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έχουμε επανειλημμένα δει να και θα τολμούσα να πω και να χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά χαρτιά ζητήματα που άπτονται αποκλειστικά τον κανονισμό της πολιτικής συνοχής και υπόκεινται σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας στην διαδικασία της συναπόφασης. Είναι λογικό αυτές οι εξελίξεις να γίνουν τις ανησυχίες μας, τόσο της Επιτροπής μας, αλλά και του πλήρου του Κοινοβουλίου. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη σας επ' αυτού του ζητήματος και πώς σκοπεύετε να το χειριστείτε. Σας εύχομαι τέλος ολόψυχα καλή επιτυχία σε αυτό το απαιτητικό έργο που έχετε αναλάβει μια και, η επιτυχία στο έργο σας για την πολιτική συνοχή θα είναι επιτυχία όχι μόνο της Ιρλανδικής Προεδρίας αλλά όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των φιλελευθέρων, κύριος Κάλαχερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον Brendan Χάουλι που είμαστε συνάδελφοι επί σειρά ετών στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και τον σέβομαι απεριόριστα. Χαίρομαι πολύ που ήρθε σήμερα για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και όπως είπε, η περιφερειακή ανάπτυξη, η συνοχή, η αναπόσπαστο κομμάτι της, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και ε, για την ανάπτυξη της μας της χώρας. Και θέλω να πω ότι ιδίω στην περιφέρεια που εκπροσωπώ, φανταστείτε, δείτε το χάρτη της Ιρλανδίας, αν δείτε τη δική μου επαρχία, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η Αλάσκα της Ιρλανδίας. Από τη μια έχει τον Ατλαντικό και από την άλλη έχουμε τη Βόρεια Ιρλανδία ε, είμαστε μια δημοκρατία ε, από μόνοι μας, αν θέλετε, ένα δικό μας κράτος, ξεχωριστό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, αναφερθήκατε και στην ειρηνευτική διαδικασία. Ήμουν βουλευτής όταν ανακοινώθηκε η καταποστηρώση και χειρία και τότε ο Ζακ Ντελόρ, πρόεδρος της Κομισιόν, είχε χαιρετήσει την ε, αγγελία αυτή και είχε πει ότι η Ευρώπη θα ανταποκριθεί θετικά και πρακτικά. Και βέβαια η Ευρώπη κατάρτισε προγράμματα. Αυτό ε, είχε, χρειαζόταν κάποιο χρόνιο, χρόνο. Αλλά η άμεση αντίδραση ήταν ότι αυξήθηκε η συμμετοχή της ε, χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ταμείο της Στήριξη της Ιρλανδίας που είχε δημιουργηθεί τη δεκαετία του 70 και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην όλη επιτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ήταν πολύ σημαντικό ότι με τη στήριξη, την πλήρη στήριξη του, του Κοινοβουλίου που απαιτεί το, αλλά δόθη ομόφωνα, κατάφερε λοιπόν η Κομισιόν να, στήριξει τόσο πολύ αυτό το ειρηνευτικό πρόγραμμα. Δεν ήταν το ίντερνετ, γιατί έτσι νομίζαμε από ε, διαμαρτυρίες. Όλα τα ασφάλματα του παρελθόντος μας έχουν διδάξει πολλά. Και άλλη πρόσθετη χρηματοδότηση χρειάστηκε. Τώρα, ε, αν δει κανεί τα τελευταία 7 χρόνια, το 2007 το 2013, 275 εκατομμύρια έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ειρηνευτικό Ταμείο. Και όταν ε, μίλησε και ο Πρωθυπουργό ε, στο κοινοβούλιο πριν εβδομάδα, μίλησε για την ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό το ειρηνευτικό ταμείο που το λέγεται PIS 3, ε, να γίνει και PIS 4, PIS 4. Και να σας πω επίσης ότι η παλιότερη περιοχή μας στην Κιλανδία ήταν στο στόχο 1 μεταξύ ε, Δύσης ε, και ενδοχώρας, κεντρικής ενδοχώρας. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει με την περιοχή μου και αν θα παίρνουμε πόρους και στη συνέχεια, αλλά ανησυχούμε, ανησυχούμε για τη λόγω των επενδύσεων που έγινε στις αρχές του 2000, πλέον η περιοχή μας θεωρείται πιο ανεπτυγμένη. Αλλά δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ για το πλατή κοινό, για τον πληθυσμό της περιοχής εκτός από τις υποδομές, που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι ανεπτυγμένη περιοχή και δεν είναι για μας θετικό γιατί το κατακεφαλήν ΑΕΠ μας είναι πάνω του 90% του μέσου όρου των 27 χωρών και αυτό χρησιμοποιείται, είναι ξέρετε ότι είναι ο δείκτης για να χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση, την κατάταξη των περιφέρειων. Δεν είναι όμως το μόνο κριτήριο, πρέπει να δείτε την απασχόληση. Ότι έχουμε 16,5% ανεργία στην Ιρλανδία και 20% κάτω του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου είναι ο μέσος όρος απασχόλησης στην περιοχή μας. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν κύριε Χάουλεν να επιχειρηματολογήσετε και να φροντίσετε στο πολιτές μεσονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 να ληφθεί υπόψη και δεν το λέω γιατί θέλω να τη δική μου μόνο περιφέρεια. Μιλάμε για πολλέ περιφέρειε. Πολλοί σαν μπορούν να αναφέρουν πάρα πολλέ άλλε περιφέρειε. Είμαι βέβαιο από διάφορε χώρε που πλήττονται από την οικονομική ύφεση και την μεγάλη ανεργία. Επειδή λοιπόν γίνεται αυτή η επανακατηγοριοποίηση με τον αδειάση των ανθρωπικών ταμείων. Ε, για την Ευρώπη ε, ουσιαστικά μιλάμε. Και βλέπουμε και κάποια προηγούμενα. Και υπάρχουν προηγούμενα. Αν δει κανεί παραδείγματο χάρη το 2007-2014. Περιφέρειες σε 20 χώρες που εγκρίθηκαν για ε, περαιτέρω χρηματοδότηση, ενίσχυση ή τέλο πάντων συμπερίληψαν σε ένα ειδικό ταμείο. Και ελπίζω να συνεχίσετε να βοηθάτε στο να αναπτυχθεί αυτή η απόκεντρη περιφέρεια της Ιρλανδίας αλλά και άλλων βέβαια περιφερειών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να τιμωρηθούμε λόγω της περίοδου αναφοράς 2007-2009, η κατάσταση δεν είναι τόσο ρόδινη ε, όσο μπορεί κάποιον θέλουν να την παρουσιάσουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ αυτό να το έχετε υπόψη σας και σας διαβεβαιώνω ότι θα έχετε τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας σας Ελπίζω να είναι άκρο επιτυχη όπω ήταν και οι έξι προηγούμενε προεδρίε. Ο Υπουργό Χάλουν και οι συνάδελφοί του είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσουν να στεφθεί και αυτή η προεδρία με επιτυχία όπω οι προηγούμενες. ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον Υπουργό αν θέλει να απαντήσει τώρα σε αυτά τα σχόλια. Σα ευχαριστώ πράγματι πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως να ξεκινήσω καλύτερα ευχαριστώντα τον κύριο Φανίστερ Ρόι για μια πολύ θετική προσέγγιση από πλευρά του και μια στεναρή αποφασιστική προσέγγιση αναγνωρίζοντας τα εμπόδια όσον αφορά την θέσπιση της ενός χρονορίζοντα όσον αφορά την ημερήσια διάταξη που θέσαμε. Δεν θα σχολιάσω το θέμα του κυρίου Κάμερον. Είναι προφανώς όλοι με πάρα πολύ προσοχή ακούμε και ακούσαμε τα όσα αναφέρονται από τον ίδιο τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αλλά για αυτά τα κονδύλια έχουν τεράστια σημασία και έχουν α, νέες, ας το πω έτσι, νέους στόχους ε, από την ε, αρχική ιδέα ότι είναι ένα ταμείο επενδύσεων, επενδυτικό ταμείο αυτή η δραστηριοποίηση. Είναι μια σημαντική ιδέα αυτή. Δεν είναι ανακατανομή κονδυλίων, είναι κονδύλια για συγκεκριμένο δεσμευτικό στόχο. Ο στόχος αυτός είναι η ανάκαμψη, η ανάπτυξη, η θέση απασχόλησης. Το να υπερβούμε τις ανισότητες που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των δράσεων. Και υποπροσωπική ε, προσέγγιση, λέω, είναι άποψή μου, όχι μόνο οικονομικά είναι σημαντικό, αλλά και πολιτικά πολύ σημαντικό. Ο πυρήνας, η καρδιά, η ιδέα της συνοχής το να εργαστούμε, να πετύχουμε κοινέ διατάξεις και προδιαγραφές ε, διαβίωσης ε, δεν είναι μικρή σημασία ε, και γι' αυτό πλήρως αναγνωρίζω και συμφωνώ με αυτό που είπε σχετικά με αυτό το θέμα ο κύριος Φανίστερ Ρόι. Σε σχέση με την πρόοδο για συμφωνίες, έχει υπάρξει πρόοδος μέχρι τώρα. Πολλές αν όχι όλες οι κυβερνήσεις εργάζονται σε ατομικά, ε, εξειδικευμένα προγράμματα από πλευρά του, προγράμματα των χωρών του. Και έτσι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, τα χρήματα των φορολογουμένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι. Οι λεπτομέρειε θα πρέπει να καθοριστούν. Η γενικότερη δομή όμω είναι γνωστή και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δράσουμε. Και υπό του όρου τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη ερώτηση που έθεσε ο κύριο Φανίστερ Ρόι για το την εργαλειοθήκη, ε, το κουτί MFF και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο έντονα αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο εξεβονίμων εδώ, τον κύριο Σταυρακάκη δηλαδή, σε σχέση με το πώς εμείς υπό το πρίσμα του Συμβουλίου θα θέλαμε να δούμε αυτά τα θέματα να προάγονται και να σημειωθεί πρόοδος. Θα ήθελα να σας διασφαλίσω σε σχέση με αυτό και προφανώς βέβαια ελβελπιστούμε ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το MFF στη συνάντηση του Συμβουλίου τώρα, αλλά και υπάρχουν και ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να είναι η πιθανή έκβαση από πλευράς του Συμβουλίου και γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος ο του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενεργά εμπλέκεται με όλους τους συμμετέχοντες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και ο Τίσοκ, ο Πρωθυπουργό μας, θα συναντήσει και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ώστε ήδη στι αρχέ Φεβρουαρίου να προλιανθεί το έδαφο ώστε να υπάρξει τελικά συμφωνία. Βέβαια το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη δική του έγκριση από πλευρά του, να συνενέσει. Και εγώ προσωπικά τι λέω. Λέω ότι η προηγούμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου κατέστησε σαφέ ο άμεσα προηγούμενος προεδρεύων του Συμβουλίου Κύπριος Υπουργό, που βρισκόταν στη θέση που βρίσκομαι εγώ τώρα διαβεβαίωσε ότι η προσέγγιση είναι αυτή όπως είναι και της Ιρλανδικής Προεδρίας και θα ήθελα εδώ να εκφράσω και με επιφύλαξη. Ξέρω ότι κάποιοι θα ήθελαν να πούν ότι ίσως μια καθυστέρηση με τον έναν ή άλλο τρόπο θα μπορούσε να διεύρυνε, λέει, τι προοπτικέ να πετύχουμε κάτι περισσότερο όσον αφορά τα θέματα συνοχή. Κρούω κόδωνα κινδύνου να μην υιοθετήσουμε μια τέτοια προσέγγιση. Δεν θα είναι αυτό επικοδομητικό. Όταν θα έχει καθοριστεί αυτό το πακέτο μέτρων λοιπόν πρώτα, μετά στη συνέχεια οι λεπτομέρειε των νομοθετικών αυτών προτάσεων θα πρέπει να επανέλθουν εδώ με τι προ... κανονικές προτάσεις για τη συνέχιση του κανονικού νομοθετικού έργου από πλευρά Ευρωβουλή. Το Ευρωκοινοβούλιο τι θα κάνει Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει αυτό. Στεναρά θα συνεργαστεί, θα εργαστεί ο συνομοθέτης διαμορφώνοντας αυτές τις προτάσεις τι οποίες θα αποστείλει πάλι προς το Συμβούλιο. Αυτή είναι η δουλειά. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση και θα συνεχιστεί έτσι η διεργασία ώστε οι απόψει του Συμβουλίου και οι απόψει του Ευρωκοινοβουλίου να μπορέσουν, α το πω έτσι, να εξεταστούν και να σφυριλατηθούν με την προοπτική να υπάρξει μια συμφωνία ώστε να μπορέσουν να πατήσουν το κουμπί του χρόνου και να έχουν συγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία θα είναι έτοιμα να δρομολογηθούν και να λειτουργήσουν. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη παρατήρηση για τη συνέργεια, απόλυτα δεν δεκτή αυτή την παρατήρηση και όπως και ο συνάδελφος Υπουργό Σέρλοκ ε, που εμπλεκόμεθα στο πρόγραμμα για τον ορίζοντα της στρατηγικής για το 2020 υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης τελικά. Να παραμείνουμε εμείς ως Ευρώπη, ως Ευρωπαίοι στο επίκεντρο της ε, καινοτομίας παγκόσμια και από πλευράς ε, Επιτρόπου Κουίν όλα αυτά και οι συνέργειες αυτές πρέπει να είναι σεβαστές. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα ισόρροπο πακέτο και αυτό είναι μέρος ε, του διαλόγου και των διαβουλεύσεων που θα πρέπει να αναπτύξουμε για να πετύχουμε αυτόν τον τελικό στόχο. Τώρα η πολιτική συνέπεια και συνεκτικότητα ως παρατήρηση του κυρίου Σταυρακάκη απόλυτα γίνεται δεκτή και τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και για τις του για επιτυχία κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Σε σχέση τώρα με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον κύριο Γκάλαχερ από την Ιρλανδία, με τον οποίο συνεργάστηκα και είναι εξέχον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στην Ιρλανδία και εξέχον υπουργό στο παρελθόν στην ε, Ιρλανδία, με συγκεκριμένε εξειδικευμένε γνώσει για τα θέματα αλληλεία. Είναι σε σχέση με αυτά και σε σχέση με την, τον Ντόνεγκαλ που βρίσκεται πιο μακριά από την δική μου περιφέρεια, βρισκόμαστε στα δύο αντιδιαμετρικά, θα έλεγα πιο απομακρυσμένα τμήματα της Ιρλανδίας θα ήθελα να αναγνωρίσω τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε η πολιτική για τη συνοχή στη χρηματοδότηση που είχε προηγηθεί ώστε σημαντικά να αλλάξει το τοπίο περιφερειακών τέτοιων επαρχιών και ε, περιφερειών όπως την δική του και αυτό ακριβώς είναι η δουλειά που ε, έχουμε αναλάβει και έχουμε επομιστεί και πρέπει να συνεχιστεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα να διαβιβαστεί και να γίνει κατανοητό. Δεν σταματάμε, δεν χαρώνουμε, Συνεχίζουμε την προσπάθεια υπέρ και προς την ε, συνεκτικότητα και συνοχή υπό όλους τους όρους και πολιτικά και οικονομικά και υπό όλες ε, τις πτυχές πολύ σχηδός. Δύο συγκεκριμένα τώρα θέματα σχετικά με την παρέμβαση του κυρίου Γκάλαχερ. Αναφέρθηκε στην ειρηνευτική διαδικασία ο κύριος Γκάλαχερ. Τώρα, σε σχέση με αυτό θα ήθελα να αναγνωρίσω την μοναδική συνεισφορά που επετεύχθη από πλευράς Ευρώπης για την σταθεροποίηση κατά το παρελθόν της ειρήνης, την εδραίωση και παγίωση της ειρήνης στην Ιρλανδία, στην Βόρεια Ιρλανδία και σε σχέση με ε, την Επιτροπή. Από πλευράς Επιτρόπου Χάν θα υπάρξει μια επίσημη εκδήλωση για την αναγνώριση αυτής της σα. και εσείς κυρία Πρόεδρε που ε, θα είσαστε προσκεκλημένοι και ελπίζω ότι θα παραστείτε και θα είσαστε και εσείς παρόντες διότι είναι σημαντικό αυτό το έργο για την συνοχή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα διαμεθοριακά, διασυνοριακά, διαπολιτιστικά, δια κοινοτικά όσον αφορά τις κοινωνίες των διαφορετικών κοινοτήτων και έτσι από πλευρά ε, ε, ε, ανώτατων αξιωματούχων, πρωθυπουργού και αναπληρωτή πρωθυπουργού και από τη Βόρεια Ιρλανδία θα υπάρξει συμμετοχή. Και τώρα, εδώ από πλευράς Προεδρίας δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο για μια συγκεκριμένη περιφέρεια της Ιρλανδίας. Όμως νομίζω ότι ένα πάρα πολύ σωστό και ορθό σημείο αναφέρατε, δηλαδή τις μεταβατικές αυτές περιφέρειες σε μια ιδιαίτερη περίοδο οικονομικής ε, δυσχέρειας όσον αφορά τη συγκυρία μας. Μια εικόνα που δίνεται σε σχέση με μια περιφέρεια που μπορεί να μην ανταποκρίνεται σωστά προς τα πράγματα. Είχαμε μια εξέλιξη που γραμμικά μπορούσε να προβλεφθεί ότι θα συνεχιζόταν. Και τώρα κάτι τέτοιο δεν ε, είναι δεδομένο. Και υποσυζήτηση βρίσκεται το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει και απόψει στο Κοινοβούλιο σχετικά. Θα υπάρξουν κάποιες περιφέρειες που για ένα χρονικό διάστημα που σε σχέση με αυτή την στιγμιαία φωτογραφία, ως στιγμιότυπο snapshot που έχουμε ενώπιόν μας, μπορεί να ε, υπάρχει κάποια δυνατότητα να επανεξετάσουμε τα πράγματα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ομαλή αυτή πρόοδος θα μπορέσει να συνεχιστεί και να τύχει, ε, ας το πω έτσι, μετεξέλιξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αλφόνς έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε της Ιρλανδίας, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι η ομάδα των Πρασίνων πρέπει να τονίσει ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την Προεδρία σας, πόσο μάλλον που σύμβολο της χώρας σας είναι το πράσινο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, πιστεύω, και ένας πολύ καλός ιονός για την Προεδρία σας. Πρέπει να πω ότι μετά από αυτά τα οποία είπατε και μετά τον λόγο σας που άκουσα και στο Στρασβούργο, καθώς επίσης και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργό σας, θεωρώ πραγματικά ότι έχετε μία βεβαιωμένη πλέον ευρωπαϊκή ευαισθησία και πραγματικά ενδιαφέρεστε για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Υπάρχει μια έντονη πολιτική βούληση και εμεί συμμεριζόμαστε πραγματικά την στάση σας αυτή στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ζωτικότητα, αυτή η αισιοδοξία την οποία εκπροσωπείτε και την οποία ακούμε κάθε φορά στις, στους λόγους στους οποίους εκφωνείτε. Πιο συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα της ε, δικής μας Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα προβληματικές και παρασκηνιακά έχουμε ακούσει ότι τα πράγματα ακόμα και να γίνουν πιο δύσκολα στην επόμενη σύνοδο σε σχέση με τα όσα έχουν ήδη γίνει στα πλαίσια του Συμβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής αυτό το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και είναι θεμελιώδες είναι η νέα αρτεκτονική η οποία έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις λεγόμενες ενδιάμεσες περιφέρειες. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη πολιτική συνοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε στην πολιτική αυτή την απαραίτητη ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τις περιφέρειες εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες περιφέρειες να μην βρεθούν εντελώ εκτεθειμένε στον ανταγωνισμό που δημιουργείται με τα μεγάλα αστικά κέντρα και με τις μεγάλες πλούσιες περιφέρειες, οι οποίε προφανώ έχουν πολύ περισσότερα οικονομικά προνόμια σε σχέση με τις μικρές περιφέρειες. Η συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά και την οποία εμείς πρέπει να προωθήσουμε. Επίσης, εσείς είπατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε όλος ιδιαιτέρως με τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες. Όντως υπάρχουν δομικές αδυναμίες για τις περιοχές αυτές. Ξέρετε ότι ε, οι πιο μονομένες περιφέρειες θα πρέπει να χαίρουν συνεχών διορθωτικών μηχανισμών προκειμένου οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης, οπουδήποτε και να βρίσκεται, σε μια πιο κεντρική ή πιο μακρισμένη περιφέρεια, να μπορεί να νιώθει ότι είναι ένας ισότιμος πολίτης με τους άλλους και ότι τυχαίνει της ίδιας αντιμετώπισης και ότι συμμετέχει επίσης όρη στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Ιρλανδική Προεδρία και ελπίζουμε ότι θα καταφέρετε πραγματικά να συμβάλλετε στο να δοθεί μια σωστή καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καπετάνια λοιπόν, καλή τύχη. Κορνέλια Ernst. Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Εξ ονόματος ε, του δικού μας συντονιστή, του κύριου Σομάτζη, που δεν μπορεί να είναι παρόν, δεν μπορεί να παραστεί, και της ε, ε, κοινοβουλευτικής ομάδας μας να σας χαιρετήσω θερμά για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Χαίρομαι ότι ανήκετε στους φίλο ευ Ευρωπαίους. Είναι σπάνιο να βρίσκει και να συναντά κανείς ανθρώπους που έχει τέτοιες θέσεις. Όλο και λιγότεροι γίνονται δυστυχώς στην Ευρώπη και αυτό δεν μας ε, ευχαριστεί ιδιαίτερα. Όμως παρόλα αυτά, τρεις παρατηρήσεις έχω. Το πρώτο είναι φυσικά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σχεδιασμού. Ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες και αν δει κανείς τις διαβουλεύσεις σε σχέση με το Συμβούλιο, τι διαπιστώνει κανείς, ότι εδώ υπάρχει ε, αντιπαράθεση, πληστηριασμός στον αγώνα για την περικοπή κονδυλίων. Εξαρτώνται όμως τόσα πολλά από αυτά τα κονδύλια και όλοι ξέρουμε θα έρθουν και άλλα κράτη που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή αυτή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωση, Πρέπει κονδύλια να διασφαλιστούν. Ερωτώ, ποια είναι η θέση της Ιρλανδίας μια και αναμένονται περαιτέρω περικοπέ από πλευρά Ιρλανδία. Η Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε μια συνέντευξη τύπου μέσων Ιανουαρίου είπε ότι 15 με 20 δι από πλευρά κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού θα περικοπούν, λέει. Με ποια διατύπωση το είπε, είπε είμαστε αρκετά πραγματιστέ και πρέπει να συμβεί αυτή, να ληφθεί υπόψη αυτή η περικοπή. Λοιπόν, ερωτώ, ποια είναι η θέση τη Ιρλανδία στι περικοπέ αυτέ, για τι περικοπέ αυτέ. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια. Πώ θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Θα συμμετάσχετε στον ανταγωνισμό πληστηριασμού για περικοπές ή θα υποβάλλετε διαφορετικές προτάσεις. Δεύτερο θέμα. Και εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια που δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια. Παρότι προέρχομαι από την πλούσια εντό εισαγωγικών Γερμανία. Έχουμε όμω διαφορετικές περιφέρειες και στην πλούσια χώρα μα. Προέρχομαι από τη Σαξονία. Έχουμε και σύνορα και ε, είμαστε δίπλα στην Τσεχία και Πολωνία και έχουμε προβλήματα στην ε, χώρα, στο κρατήδιό μας, ανεργία. Είχαμε ε, υψηλό ποσοστό σε σχέση με την, ε, την αρχή της νέας χιλιετίας ως μεταβατική περιφέρεια προσωρινής κατηγορίας θα έχουμε αρνητική αντιμετώπιση. Ανησυχούμε ιδιαίτερα. Έχουμε 55 περιφέρειες που αφορώνται από αυτό το θέμα. Θα περικοπούν σημαντικά τα κονδύλια τα οποία μας δινόντουσαν. Τα ποσά. Αυτό είναι ολέθριο για μας. Οι υποδομές σε μια ολόκληρη σειρά χωρών που έχουν τέτοιες περιφέρειες μεταβατικές ή προσωρινές εξαρτώνται υποδομές από τα κονδύλια. Μπορείτε να πείτε κάτι για αυτό το πρόβλημα. Τελευταίο θέμα. Κάθε χρόνο γίνεται λόγος εκ νέου για μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης Ξέρετε, υπάρχει κίνδυνο όταν διαρκώ συζητά κανεί και αναφέρει ένα θέμα χωρί να γίνεται κάτι, αυξάνεται και δεν μειώνεται το γραφειοκρατικό βάρο στο τέλο τέλο. Κάποια πράγματα θα μπορούσαν ε, να ελαφρυνθούν όσον αφορά την γραφειοκρατική επιβάρυνση. Τι θα κάνετε εσεί ω Ιρλανδική Προεδρία για να το πετύχετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα προσεκτικά και θυμήθηκα κάτι που έγραψε ο Hans Christian Andersen ότι τίποτα το μεγάλο δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς ε, να συμμετέχει φαντασία στη δημιουργία αυτή. Μεγάλες επενδύσεις ε, σε σχέση για παράδειγμα με τις δράσεις αυτές ε, που προσήλθαν σε μας ε, μας είπαν ότι υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και γι' αυτό ε, προσήλθαν ε, αυτές οι επενδύσεις. Μπορώ να πω ότι η δική σας ενθουσιώδης αυτή προσέγγιση διαδραματίζει και αυτή ένα ρόλο. Το 2010 είχα πάει στην Ιρλανδία ως εισηγητής για τα θέματα του προϋπολογισμού και συνάντησα εκπροσώπους του Ιρλανδικού Υπουργείου Οικονομικών. Τι μου είπαν οι Ιρλανδοί εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών Επιτόπου, ότι η Ιρλανδία ωφελήθηκε και άντλησε τα περισσότερα κονδύλια και με τον καλύτερο τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ταμεία διαρωτηθήκαμε και προβληματιστήκαμε πώς τα κατάφερε αυτά η Ιρλανδία, πώς μπόρεσε να γίνει αυτό. Έχουμε διαφορετικές απόψεις εμείς. Δηλαδή, οι περιφέρειες θα πρέπει να ρυθμίζουν την άντληση αυτών των κονδυλίων από τα ταμεία ή κυβερνήσεις. Ή μήπως θα πρέπει οι τοπικές αρχές και κυβερνήσεις ε, ε, τοπικού και δημοτικού επίπεδου να το κάνουν. Εγώ ανήκα σε ένα τέτοιο τοπικό περιφερειακό όργανο. Ερώτησα τι έγινε σε εσά και μου επεξήγησαν ότι κεντρικά με κεντρικό σχεδιασμό είχε σχεδιαστεί αυτό. Όχι ε, δηλαδή από την περιφέρεια αλλά από το κέντρο. Θα έλεγα ότι τη δική σας αυτή πείρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τα κονδύλια από το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Ευχαριστώ. Uh, thank you again. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ και πάλι. Να ξεκινήσω με τον κύριο Αλφονσί. Πρώτα απ' όλα, ναι, πράγματι, το πράσινο είναι το χρώμα της Ιρλανδίας, ε, το γρασίδι μας είναι πράσινο, ε, αλλά ε, και το βοδινό μας είναι πολύ καλό. Επίσης εκφράσατε ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες συζητήσεις για το πολιτές μεσορμικό πλαίσιο. Ανέφερα ήδη τις προσδοκίες που έχουμε για τις αρχές Φεβρουαρίου. Στις 7 και 8 που συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Φον Ρομπόι νιώθει ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Προφανώς, όπως είπα, θα δώσετε κι εσείς εδώ το Κοινοβούλιο την έγκριση εν συνεχεία. Και το σημαντικό είναι η ουσία των ε, συνιστοσών του διαπραγματευτικού κουτιού για το πολιτισμό οικονομικό πλαίσιο. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα έχουμε ένα καλό πακέτο μέτρων για τη συνοχή. Γιατί αυτό αποτελεί δική μου ευθύνη, είμαι επικεντρωμένο στην προσπάθεια αυτή και είμαι αισιόδοξο ότι θα το πετύχουμε. Βέβαια, τι λεπτομέρειε θα πρέπει να τι επεξεργαστούμε σε το χρόνο. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό όραμα, τον, την αισιοδοξία, εγώ είμαι αισιόδοξο και η Ιρλανδία είναι αισιόδοξη χώρα. Παρότι έχει περάσει ίσως στη δυσκολότερη της περίοδο τα τελευταία τρία χρόνια. Στην διάρκεια του πολιτικού μου βίου τουλάχιστον αυτά ήταν τα πιο δύσκολα τρία χρόνια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε και τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η ανάπτυξη και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο για το μέλλον, το οποίο θα βασίζεται όχι στις τράπεζες και στην κερδοσκοπία, αλλά στην καινοτομία, στις εξαγωγές, και πραγματικά είμαστε σε καλό δρόμο να το πετύχουμε. Δεν θέλω να καταχραστώ τις θέσεις μας προεδρεύοντος ε, και να πω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια, γιατί όμως πράγματι χρειαζόμαστε, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, να μεταλαμπαδεύσουμε το, την αισιοδοξία μας για το μέλλον της Ιρλανδίας και σε μια αισιοδοξία για το μέλλον της Ευρώπης, παρότι υπάρχουν κάποιες ε, φωνές που εκφράζουν διαφορετικά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το ευρωπαϊκό Ρώμα είναι το πιο πολύτιμο και σημαντικότερο project που έχει ποτέ αναλυφθεί στην Ευρώπη. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό για κάποιες ε, ενδιάμεσες, ε, αν θέλετε, περιφέρειες και μιλήσατε για τους ε, απορροφητές κραδασμών, τέλος πάντων σαν προφυλακτήρες, κάτι τέτοιο. Και ήταν πολύ ωραία, εύστοχη αυτή η παρομοίωση. Το θέμα να μην μείνει κανένας πίσω. Και σίγουρα πρέπει να βρούμε και συμπληρωματικά εργαλεία για να το πετύχουμε. Αυτό βέβαια είναι η δουλειά των ε, δημοκρατικά εκλεγμένων ε, βουλευτών, άρα ημών των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές ε, περιφέρειες για τις οποίες μιλήσατε, άκουσα αυτό που είπατε. Η Ιρλανδία, η δική μου χώρα, περιγράφεται σαν νησί ενός νησιού μιας υπήρου είναι περιφερειακή χώρα και σίγουρα οι περιφερειακές περιφέρειες, οι απόκεντρες περιφέρειες αναφέρονται συγκεκριμένα, γιατί δική μου σε αυτές, στη συνθήκη. Και επομένως πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο συζητήσουμε. Την κυρία Ένστ, που και αυτή εξέφρασε κάποιες ανησυχίες για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και συγκεκριμένα είπε ποια είναι η Ιρλανδική θέση. Αυτή ήταν η ερώτησή της. Θα μπορούσα να σα πω το εξή. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, ε, παραφράζοντας τον, είπε ότι η Ιρλανδία θέλει μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σωστή χρηματοδότηση που να λειτουργεί σωστά, με το σωστό μείγμα προτεραιοτήτων, με δίκαιη κατανομή των πόρων και με επίκεντρο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει έναν προπολογισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί στο στόχο αυτό. Και αυτό θα είναι και το δικό μα καθήκον στη διάρκεια τη Ιρλανδική Προεδρία. Και ελπίζουμε στο βαθμό του δυνατού να το πετύχουμε. Γιατί βέβαια δεν είμαστε παρά μία από τις 27 χώρες παρότι ασκούμε την Πρόεδρε αυτό το εξάμεινο. Άμεσα, άμεσα, όχι στο απότερο μέλλον, θέλουμε να εξασφαλίσουμε έναν προπολογισμό που να είναι ο κατάλληλος για τους στόχους που έχουμε θέσει. Αντιλαμβάνομαι επίσης ε, αυτό που είπατε για φτωχές περιφέρειες, φτωχές περιοχέ μέσα σε πλούσιες χώρες πολλές φορές μπορεί να κατηγοριοποιήσουμε ολόκληρες χώρες και αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος ε, περιφερειών που είναι σε υπονεκτική θέση ή κάποιων πληθυσμών για ιστορικούς λόγους μέσα σε κάποιες περιφέρειες περιφέρειες, μέσα σε κάποιες χώρες. Και είπατε επίσης ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρξει απλούστευση. Το είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου. Δημιουργήσαμε ένα νέο Υπουργείο στην Ιρλανδία, το δικό μου συγκεκριμένο Υπουργείο. Εγώ είμαι Υπουργό Δημοσίων Δαπανών Άρα είμαι αρμόδιο για όλε τι δημόσιες δαπάνε. Αλλά είμαι και υπουργό μεταρρύθμισης. Διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο παρέχονται οι δημόσιες υπηρεσίες για να μπορούν να επιτελούν το στόχο τους, να υπηρετούν το σκοπό τους, για να μην έχουμε απώλειες. Και τα χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να πηγαίνουν στις ανάγκες, να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου. Και αυτά τα οποία γίνονταν πριν από 50 χρόνια δεν πρέπει να συνεχίσουμε να τα κάνουμε τον ίδιο τρόπο επειδή πάντα έτσι γινόταν. Αυτό λοιπόν το επίπεδο απλούστευσης και μείωσης της γραφειοκρατίας είναι σίγουρα σημαντικό για εμάς. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε και τις νομικές δομές και υποχρεώσεις και να υπάρχει βέβαια και ευθύνη, λογοδοσία. Για τον κύριο Μάνκα Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Μάνκα, για το σχόλιο που κάνετε σε σχέση με το πάθος. Ελπίζω να το νιώσατε ότι πραγματικά ε, δεν κατεχόμαστε από πάθος και τώρα κατά πόσον θα πρέπει να είναι κεντρική ή περιφερειακή η διάθρωση. Αυτό θα πρέπει να το δουν τα κράτη-μέλη γιατί η κλίμακα είναι σημαντικό πράγμα και εγώ έχω την εμπειρία μόνο στο δικό μου, το νησί, την Ιρλανδία. Εμείς βλέπουμε το Νότο και την ε, Ανατολή είναι πιο ανεπτυγμένη περιοχή, αλλά και στο κέντρο και στη Δύση ε, πιο υποβαθμισμένη, αλλά και μεταξύ αυτών υπάρχουν ε, διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές περιοχές και θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και διάρθρωση. Να συντονίζουμε τα πράγματα με καλό τρόπο. Μιλάω για την Ιρλανδία φυσικά και αυτό που λειτουργήσε πολύ καλά είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα το αποφασίσουν όμως, ε, τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τέσσερι έχω στον κατάλογο. Να μου πείτε, άλλοι θα παρέμβουν, αλλιώ κλείνει ο κατάλογο και θα ξέρουμε πώ θα διαμορφώσουμε το χρόνο τη ε, συνάντησή μα, τη συνεδρίασή μα. Πέντε λοιπόν είναι οι αγορητέ. Ίσως οι πέντε να ομαδοποιηθούν στις παρεμβάσει του, Ο κύριος Μποστινάρου έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είχα το προνόμιο να σας συναντήσω πέρυσι και <clears throat> συνάντησα επανειλημμένα τους συναδέρφους σας, τους υπαλλήλους σας και πρέπει να πω Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με αυτή τη συνεργασία μαζί τους και τις θεσμικές σχέσεις που θεσπίσαμε και θεσμοθετήσαμε. Η Ιρλανδική Προεδρία ξεκινά καθώς εορτάζει η Ευρώπη τα 50 χρόνια της συνθήκης γερμανογαλλικής συνθήκης ε, των ηλισίων. Είδα στην τηλεόραση μία επισκόπηση, μία αναδρομή των σχέσεων Ντεγκόλ και Άντεναουερ με αυτή τη συνθήκη. Και βλέπουμε ότι σε περίοδο κρίσης χρειαζόμαστε περισσότερο από οποτεδήποτε όχι μόνο δεσμεύσεις και οράματα αλλά επίσης υψηλέ φιλοδοξίες για την δική μας αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακριβώς αυτά, αυτά τα οποία μας είπατε εσείς, αυτά τα οποία μας λέτε και αυτά που ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός είπε προσφωνώντας την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, περίοδο συνόδου της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι αυτά καλοδεχούμενα, γιατί όχι μόνο δείχνουν ότι είναι στεναρά και είναι δεσμευτικά, αλλά κάνουν, εκφράζουν μια χώρα που ωφελήθηκε από την πολιτική συνοχή. Έχετε κάθε δικαίωμα εσείς. Έχετε δικαίωμα να πείτε ότι χωρίς αυτή την ε, πολιτική συνοχή και χωρίς την βοήθεια δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Και αυτό επειδή στο Συμβούλιο ακριβώς είναι η μάχη που δίνεται, η κονίστρα, το πεδίο ε, που πρέπει αυτά τα θέματα να εξετάζονται. Η πολιτική, για παράδειγμα, ε, περικοπών κονδυλίων, λιτότητας, έναντι της ε, Ευρώπης των 27, συν ενός δηλαδή 28 με τη διεύρυνση, Πρέπει να δούμε, θα γίνουν τέτοιου είδους περικοπές ή θα συνεχίσουμε την προηγούμενη πολιτική. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συζητήσεις που είχα κατά το παρελθόν με τους αξιωματούχους σας, οι τριμερείς διάλογοι υπό την ιδιότητά μου ως εισηγητού για το Ταμείο Συνοχής, οι τριμερείς διάλογοι θα είναι πολύ καλά προπαρασκευασμένοι θα είναι μια σύντομη και πολύ καλά επικεντρωμένη, εστιασμένη συζήτηση και διαβούλευση στη διαπραγμάτευση και στο τέλος θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι το οποίο ακριβώς χρειαζόμαστε. Νομοθετικό έργο που έγκαιρα θα έρθει και που θα είναι καλά προετοιμασμένο και καταρτισμένο, σχεδιασμένο ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης και δράσης ώστε πολιτική συνοχή να μπορέσει να λειτουργήσει όπω πρέπει ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2014. Επανειλημμένα όπω αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο Μάρτιν Σούλτ του Ευρωκοινοβουλίου και από του πιο σημαντικού ομιλητέ για τα θέματα προϋπολογισμού και τα πιο σημαντικά θέματα τομεακών πολιτικών στην Ευρώπη αυτό αναφέρθηκε και στο Ευρωκοινοβούλιο και εκτό. ότι κανένα προπολογισμό δεν θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κανένα συμβιβασμό δεν θα γίνει δεκτό και δεν θα εγκριθεί αν εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορέσουμε να διαβουλευθούμε Διαφορετικά θα απορρίψουμε, λαμβάνοντα υπόψη αυτά που είπατε πιο πριν. Η Ιρλανδική Προεδρία θα έρθει δίπλα ο σύμμαχος στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι για να απορρίψει, γιατί η βούλησή μα δεν είναι να απορριφθεί το ε, σχέδιο για το, EM, ε, για το ε, MFF, αυτό θα ήταν ευθυνό πολιτικό τέχνασμα. Για να κερδίσουμε την πολιτική μάχη. Θα, μας, θα ενωθεί σε εμά ω Ευρωκοινοβούλιο η Ιρλανδική Προεδρία για, αυτή τη σημαντική μάχη για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Εσείς κύριε Νίκο Χρυσόγελ έχετε τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια εποχή κρίσης και είναι σύμπτωση ότι ξεκινώντας από την Κυπριακή Προεδρία μέχρι και τις ευρωεκλογέ, την Προεδρία θα την έχουν χώρε που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν ζήσει την κρίση και άρα ξέρουν ότι απαιτούνται πολιτικές εξόδου από την κρίση ισορροπημένες. Είναι σημαντικό να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρώπη δεν είναι καλή μόνο στην περίοδο της ευημερίας της οικονομίας αλλά και σε περίοδους κρίσης γιατί μπορεί να αλλάζει και να προσαρμόζει τις πολιτικές της ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα τον, ε, τον Μάιο του 2014 στις ευρωεκλογέ. Δεν θα μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Και νομίζω ότι όλοι εδώ μέσα μας ενδιαφέρει να διατίθενται οι ευρωπαϊκοί πόροι με αποτελεσματικότητα, το best spending που συζητάμε. Αλλά τι σημαίνει καλύτερη διάθεση των πόρων. Σημαίνει αφενός να χρησιμοποιηθεί σωστά ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υλοποιηθούν οι πολιτικές οι οποίες αφασίζουμε. Αλλιώς αν δεν υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα λέμε εδώ πέρα μόνο ευχές και το δεύτερο είναι να είναι δίκαιος ο προπολογισμό. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης δεν μπορούμε να μειώνουμε τον προπολογισμό, τον ευρωπαϊκό, που είναι έτσι καλλιώς μικρός, πρέπει να αυξηθεί και με ίδιους πόρους και φυσικά να πετύχουμε και στις πολιτικές που έχουμε θέσει στο Ευρώπη 2020. Να μειωθεί η φτώχεια, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν οι νέοι σήμερα. Εφαρμόστηκε για μια μεγάλη περίοδο πολιτική λιτότητα σε πολλέ χώρε εκ των υστέρων βλέπουμε ότι και ο ε, και ο σχεδιασμός ήταν λάθος. Υπάρχουν πολύ σημαντικές εκθέσεις και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Κομισιόν που δείχνουν ότι η λιτότητα όπως εφαρμόστηκε δεν οδηγεί σε αντιμετώπιση και των δημοσιονομικών προβλημάτων. Αυτό το έχουμε ζήσει πολύ έντονα στην Ελλάδα. Δηλαδή όσο εντείνεται η πολιτική λιτότητα τόσο αυξάνονται τα δημοσιονομικά προβλήματα. Ένα νούμερο θα σας πω. Τα μέτρα του καινούργιου μνημονίου είναι 13,5 δισεκατομμύρια και μέσα στο 2012 οι πολίτες έχουν ε, χρέος προς το δημόσιο το ίδιο ποσό. Δηλαδή, ό,τι αφαιρείται με τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και της κοινωνικής πολιτικής, σήμερα χρωστιέται από τους ανθρώπους, από τους πολίτες, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν πλέον. Άρα δεν έχει καν αποτέλεσμα. Πρέπει να, να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά, αλλά μέσα από τη μεταρρύθμιση οικονομίας, μέσα από καλύτερη λειτουργία της δίκης και μέσα από στοχευμένες επενδύσεις. Γι' αυτό μιλάμε εδώ για ταμεία τα οποία είναι διαρθρωτικά και επενδυτικά Δηλαδή το 80-90% του προπολογισμού του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου θα είναι επενδύσει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και την κρίση. Και είναι πολύ, σημαντικό αυτό. Να βελτιώσουμε βέβαια την επίδοση των προγραμμάτων. Να βελτιώσουμε το πώ εφαρμόζονται τα προγράμματα χρηματοδοτικά στι χώρε μέλη. Σίγουρα χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν πρέπει να μειωθεί ο προπολογισμό. Αναφέρω ένα παράδειγμα που το στάγαμε πριν λίγη ώρα εδώ στην ίδια Επιτροπή για τα προβλήματα των άπορων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατεθούν 2,5-3 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή όμως που αυξάνεται ραγδαία η φτώχεια και απαιτείται ενίσχυση και των πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και χρηματοδοτικά εργαλεία για τους ανθρώπους που είναι άποροι πλέον, που είναι άνεργοι, που δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια, έχουμε ενεργειακή φτώχεια. Και εσείς ξέρετε πολύ καλά νομίζω ότι εάν κάνουμε επενδυτική πολιτική μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα γιατί ξέρω ότι για τα θέματα των ανισοτήτων στην υγεία έχετε ένα πρόγραμμα που συνδυάζεται με επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία. Να βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέμε εδώ μέσα ότι οι επενδύσεις στην κοινωνική πολιτική, στην πολιτική συνοχή, στην περιφερειακή ανάπτυξη θα αντιμετωπίσουν πολλαπλώς προβλήματα, θα δημιουργήσουν θέσει εργασία, θα ζήσουν οι άνθρωποι καλύτερα, θα χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι επιδόματα για να επιβιώσουν. Και τέλος θέλω να σας πω κάτι επειδή είσαστε πραγματικά και νησιωτική χώρα. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις πολιτικές για τα νησιά. Είναι πολύ σημαντικό. Τα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ μικρό μέρος, μια πολύ μικρή έκταση και πολύ μικρός ε, πληθυσμός σε σχέση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο αξιών, σε επίπεδο οικονομία και στο παρελθόν έχουν παίξει ιστορικό ρόλο και το δικό σα νησί. Επομένω, πρέπει μέσα στη δικιά σα Προεδρία να αναλυθούν περισσότερε πρωτοβουλίε και για τον νησιωτικό χώρο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ρικάνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, Προεδρεύοντα για την εξαιρετική εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέργεια που προδιαγράψατε ως προοπτική και επιθυμία της Προεδρίας σας. Αυτή η συζήτηση, σε αυτή τη συζήτηση έγινε λόγος για τη σπουδαιότητα της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής για τις επενδύσεις. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που επιλέξατε αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό και το τονίσατε με αυτόν τον τρόπο και θα υποστηριχθεί έτσι η πολιτική συνοχή στις διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να κάνω λόγο για την συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ περιφερειών και διαμεθοριακά, διασυνοριακά. Έχουμε κάνει πολλές φορές λόγο για αυτό το θέμα στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και ξέρουμε ποια είναι η σπουδαιότητα να υπάρχει πρόσθετη αξία σε σχέση με αυτή την ευρωπαϊκή δράση και προσέγγιση. Και τώρα σε σχέση με τι διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο, η θέση του Ευρωκοινοβουλίου για παράδειγμα, ζητώντα ένα 7% για αυτά τα προγράμματα και σχέδια, φαίνεται ότι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο δεν είναι τόσο φιλόδοξη όσο εμεί ω Ευρωβουλή με αυτό το ποσοστό το 7% που προτείνουμε. Ποια είναι η άποψη άποψή σε σχέση με τη χρηματοδότηση λοιπόν αυτής της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών, διαπεριφερειακά. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε, θα θέλατε να υποστηρίξετε και να αυξήσετε αυτό το ποσοστό, αυτό το 3% λέει τώρα η ομιλήτρια που είχε αρχικά προταθεί σε σχέση με την Επιτροπή. Yes, Ο κύριος Γιάνν Όλμπριχτ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ πολύ για τον λόγο που μας εκφωνήσατε. Δίνει ο λόγος σας τις θετικές προοπτικές για μας. Όμως για την Ιρλανδική Προεδρία η χρονική συγκυρία δημιουργεί μια κατάσταση σε σχέση με τις προσδοκίες μας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το κυριότερο σημείο. Διαπραγματεύσεις όσον αφορά το, τη, τη δέσμη μέτρων εμείς ε, ε, προσδοκούσαμε, φυσικά δεν μπορείτε να παρουσιάσετε και να προασπίζετε ιρλανδικές απόψεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας, αλλά ως κάποιος που προέρχεται από μια χώρα από την ε, κατηγορία της ομάδας ε, Better Spending ή Friends of Cohesion δηλαδή θα ε, ελπίζαμε ότι σε σχέση με το Συμβούλιο θα μπορούσε να υπάρξει μια ας το πω έτσι διαφοροποιημένη προσέγγιση. Έχουμε πολλά ερωτήματα τα οποία δεν είναι σήμερα θέματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν. Θα υπάρξει αποσαφήνιση της κατάστασης κατά τους επόμενους μήνες μήνες σίγουρα. Όμως υπάρχουν κάποια πολύ ευαίσθητα θέματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και ελπίζω ότι εσείς θα μπορέσετε επίσης να διασφαλίσετε ότι η πολιτική συνοχή και τα στοιχεία της δεν θα αμεληθούν. Φυσικά όλα μπορούν να διαπραγματευτούν μεταξύ κρατών μελών, αλλά κάτι υπάρχει που βρίσκεται και στη δική μας αρμοδιότητα ως Ευρωβουλή και θα θέλαμε έτσι να ε, συμμεριστούμε τις δικές μας προσδοκίες μαζί σας όσον αφορά τους κινδύνους ή τις ε, προοπτικές αυτής της διαπραγμάτευσης. Χωρίς να επισέθω σε λεπτομέρειες θέλω να πω τα εξής. Αναφέρατε την Πολωνική Προεδρία. Είμαι Πολωνός και δεν είναι μόνο το επειδή υπάρχουν πολλοί Πολωνοί στην Ιρλανδία, αλλά και σε σχέση με την ε, επιρροή που μπορεί ίσω να ασκούν στην ε, ε, προσέγγιση. Η αμοιβαιότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό βέβαια. Η Πολωνική όμως Προεδρία ήταν εκείνοι που σε διαρκή επαφή με το Ευρωκοινοβούλιο με διαφανέστατο τρόπο προσπάθησε να προαγάγει τους στόχους τη. Οι υπεύθυνοι της Πολωνικής Προεδρίας ήταν παρόντες λοιπόν και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και πολύ συχνά συμμεριζόμενοι τις πληροφορίες, ε, τις αμφιβολίες, όλα τα στοιχεία για όλα αυτά. Αν μπορώ κάτι να προτείνω από πλευρά της Πολωνικής Προεδρίας σαν κληροδότημα είναι αυτή η διαφάνεια και το να συμμερίζεστε τις απόψεις και τις προτάσεις ε, εσείς ως Προεδρία μαζί μας ακόμα και αν η συγκυρία είναι δύσχερη, είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αλλά α φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία ε, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Α το προσεγγίσουμε έτσι. Πολιτικό σα σχεδιασμό ποιο είναι το πρόγραμμά σα. Να υπάρξουν τα τελικά, πακέτα, τα τελικά στοιχεία του πακέτου αυτού πριν από τι θερινέ διακοπέ που θα έχουν ρυθμιστεί για το Κοινωνικό Ταμείο, Διαθωτικό Ταμείο κατά τη διάρκεια τη Ιρλανδική Προεδρία. Κατά τη δική σα λοιπόν Προεδρία να μπορέσει αυτό να κλείσει. Έτσι θα προεδρεύσετε λοιπόν και στους τριμερείς διαλόγους ε, και στις ομάδες εργασίας. Είναι σαφέστατο το ερώτημα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με βεβαιότητα, αλλά έχετε μια τέτοια πολιτική βούληση ως σχέδιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κολάσκη παρακαλώ. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, domnule președinte, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εκτιμώ ιδιαίτερα την θετική αυτή αρχή της Ιρλανδικής Προεδρίας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Εκτιμώ επίσης πάρα πολύ τα όσα είπατε στην δική μας την Επιτροπή, ιδίως όταν είπατε ότι η Ιρλανδία θέλει πραγματικά μια καλά χρηματοδοτούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ότι θεωρείται ότι όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην πολιτική συνοχή. Το Ταμείο Συνοχή είναι όντω, όπω πολύ σωστά το είπατε, το βασικό επενδυτικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Δυστυχώ όμω. Τους τελευταίους μήνες μας φτάνουν διάφορα αρνητικά νέα για περικοπές προπολογισμού, για μέτρα λιτότητας και σημαντικές περικοπές στον ίδιο τον κοινοτικό προπολογισμό. Προέρχομαι από την Ρουμανία, μια ανατολική χώρα, μια χώρα από το πρώην Σοβιετικό μπλοκ. Είμαι κι εγώ μία, προέρχομαι από μια χώρα συνοχής. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλές απαιτήσει από το Ταμείο Συνοχής και εξαρτώμαστε πάρα πολύ από το Ταμείο αυτό, ιδίως στη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο. Αναφερθήκατε και εσείς στο μέλλον του Ταμείου Συνοχής μετά το 2013, μετά το 2030 με συγχωρείτε. Το μέλλον του Ταμείου Συνοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες σύγκλησης. γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στην χρηματοδότηση της συνοχής από τη μία και στο ότι θα πρέπει η συνοχή να αφορά όλους από την άλλη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους σας τους συναδέλφους για τις πολύ αυτές κέρυες παρατηρήσεις τις οποίες κάνανε όσον αφορά την κοινή αυτή ατζέντα που έχουμε. Κύριε Μποστινάρου, όντως κάναμε τις συζητήσεις αυτές στις οποίες αναφερθήκατε πέρυσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας τότε και όντως ε, αναφερθήκατε σε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Όντως ε, εορτάζουμε τα 50 χρόνια της συνθήκης των Ηλισίων και θα έλεγα επίσης ότι γιορτάζουμε επίσης και την 40η επέτειο προσχώρησης Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα οι τέσσερις αυτές δεκαετίες, οι οποίες όμως άλλαξαν, μεταμόρφωσαν πραγματικά την Ιρλανδία. μια χώρα η οποία εξαρτηθεί πάρα πολύ από το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, όσον αφορά τις εξαγωγέ, όσον αφορά ακόμα και τον πολιτισμό. Και μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά βοήθησε την Ιρλανδία να ανθίσει πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το θυμόμαστε. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να ζητούμε συγγνώμη επειδή έχουμε πολύ υψηλέ φιλοδοξίε. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ακόμα και δεν μπορούμε να πετύχουμε πάντα του στόχου μα. Πριν από λίγο καιρό ξαναδιάβασα του λόγου ε, των ανθρώπων που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρήκατε και γυναίκε, ρωτάει η πρόεδρος. Η Σας το λέω αυτό, αναφέρομαι στου άνδρες και στι γυναίκε που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω άνδρε, πρέπει να το παραδεχτώ. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν η έμπνευση της γενιάς εκείνης η οποία έβγαινε από τον πόλεμο, η οποία πραγματικά ταλανιζόταν από την ένδια. Χρειαζόμαστε την έμπνευση αυτή προκειμένου να καταφέρουμε να κινηθούμε στο μέλλον, στο μακρύ αυτό ταξίδι μας περιμένει. Καταγράφω λοιπόν πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μποστινάρου για την νομοθετική διαδικασία. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε οραματιστές ένας φίλος μου και συνάδελφός μου που ήταν υπουργό την τελευταία φορά που ήμουν και εγώ υπουργό, που είναι τώρα πρόεδρος όμως της ε, Ιρλανδικής Δημοκρατίας, πήγε κάποτε σε ένα συμπόσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρουσιάστηκε εκεί πέρα ως ο Ιρλανδός υπουργό της φαντασίας. Νομίζω ότι κακό δεν κάνει να έχει μια χώρα έναν υπουργό φαντασίες γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε όραμα. Χρειαζόμαστε όμως και ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο σε πρακτικούς όρου. Χρειαζόμαστε του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι πραγματικά το όραμα μπορούν να το κάνουν πράξη. Και ακριβώ στο συνδυασμό αυτό χρειαζόμαστε του επόμενου έξι μήνε. Χρειαζόμαστε δηλαδή σωστή νομοθετική διαδικασία για την συνοχή του επόμενου μήνε, η οποία όμω θα πρέπει να έρθει εγκαίρω. Να πω επίση, να αναφερθώ σε κάποια σχόλια που έκανε και ο κύριο Μποστινάρο αλλά και άλλοι συναδελφοί σα όσον αφορά τον προπολογισμό. Ποια είναι η άποψη τη Ιρλανδική Προεδρία όσον αφορά την ενδεχόμενη απόρριψη. Πρέπει να σας πω ότι περιμένω τελικά ότι τελικά θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα αμοιβαίω αποδεκτό. Ξέρετε πολλέ πολλές το να κυνηγάμε το καλύτερο μπορεί να είναι ιδιαίτερα αρνητικό στη τελευταία ανάλυση. Δεν θα μα βοηθήσει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Α προσπαθήσουμε τελικά να βρούμε μια συμβαστική λύση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία όμω δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει του πάντε α το αποδεκτούμε αυτό. Θεωρώ ότι αν απορρίψουμε την δυνατότητα μιας πρώτης συμφωνίας, αυτό δεν θα αποτελέσει καμία περίπτωση εγγύηση ότι θα έχουμε συμφωνία στο μέλλον. Ο Έλληνας συναδελφός μου, ο κύριος Χρυσόγελος, ελπίζω να, να προφέρω σωστά το επίθετό σας, Χρυσόγελο. Πρέπει να κάνω καλύτερη εξάσκηση στα ελληνικά μου. σα ζητώ συγγνώμη, λέει ο Υπουργός. Πραγματικά νομίζω, κύριε Χρυσόγελε, ότι θέσατε κάποια θεμελιώδη ερωτήματα για τους δημοκράτες. Από τη στιγμή που υπάρχουμε ως βουλευτές, υπάρχουμε μόνο για να εκφράζουμε τη βούληση των λαών, των πολιτών. Ποιο μήνυμα λοιπόν εμεί διαβιβάζουμε προ του πολίτε. Πώς μπορούμε να τους ζητάμε να μας στείλουν σε ένα θεσμικό όργανο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να επιτελέσουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν τα όσα είπατε. Και ως ε, Ιρλανδός Υπουργό Αρμόδιος για θέματα προπολογισμού, καταλαβαίνω πολύ καλύτερα από άλλους μου συναδέλφους τι σημαίνει λιτότητα. Τι σημαίνει λιτότητα όσον αφορά το ότι ταράζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στους δημοκρατικούς θεσμούς. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να μετριάσουμε την λιτότητα, την οποία δεν μπορεί να αποφύγουμε αν θέλουμε τελικά να πετύχουμε δημοσιονομική εξυγίανση και ισοσκελισμένο προπολογισμό. Χρειαζόμαστε όμω ένα μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων τη λιτότητα μέσω οικονομική ανάπτυξη, μέσω θέσεων εργασία. Και αυτόν τον διάλογο ξεκινήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν αφορά αυτό μόνο τη δική μου τη χώρα, αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καταγράφω πάρα πολύ όλα αυτά τα οποία είπατε για την Ιρλανδία. Κυρία Μάνερ. Αναφερθήκατε στην ε, πολιτική επενδύσεων, στι επενδύσεις που έχουν γίνει, αναφερθήκατε στην περιφερειακή συνεργασία και ποιο είναι το επίπεδο του προπολογισμού που ενδεχομένω να δοθεί στην περιφερειακή πολιτική. Ακούω πολύ προσεκτικά τα όσα είπατε και γνωρίζω ότι έχουν γίνει κάποιες ε, συζητήσεις. Θα δούμε ποια ήταν η έκβαση των συζητήσεων αυτών. Κατάλαβα πάντως ακριβώς τι θέλετε να πείτε και έχετε κάποια πολύ σημαντικά επιχειρήματα. Κύριε Όλμπριχτ, με ρωτήσατε ποια θα είναι η έκβαση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά το νομοθετικό αυτό πακέτο. Η δικιά μου εκτίμηση θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις αλλά για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε τη δική σας κατανόηση, ανοχή, συνεργασία, προκειμένου να καταφέρουμε από κοινού να συνεργαστούμε και να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό πακέτο το οποίο θα εγκριθεί και το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να σημειώσουν πρόοδο προς μία νέα διάρθρωση για την περιφερειακή πολιτική από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι ο ρόλος που μπορούμε να διαδραματίσουμε ως προεδρεύοντες είναι κυρίως τεχνικός. Σαφώς μπορούμε να έχουμε ένα όραμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε και από τεχνική πλευρά να προωθήσουμε τι προτάσει οποίε επεξεργαζόμαστε. Και εμεί θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είμαι σίγουρο ότι έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από την δική σα την ικανότητα, την δεξιότητα, καθώ επίση και από τα όσα κατέδειξε ω ε, εμπειρογνωμοσύνη η ε, Πολωνική Προεδρία. κύριος Ματούλα από την Ρουμανία. Ο ρόλος της συνοχής ως μέσο για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προφανώς είναι κάτι το οποίο τόνισα και εγώ πάρα πολλές φορές. Θέσατε όμως ένα δύσκολο ερώτημα όσον αφορά τις προσδοκίες. Πρέπει να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε τις προσδοκίες στην πραγματικότητα. Ξέρετε ότι είναι περιορισμένοι οι προπολογισμοί, υπάρχουν όρια, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε δυνατή ανάγκη. Δεν νομίζω λοιπόν θα πρέπει να τροφοδοτούμε προσδοκίες οι οποίες δεν είναι ρεαλιστικές. Αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Βανιστερόη, το ότι ο βασικός μας ρόλος είναι να καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο νομοθέτημα και σε τέτοιους προπολογισμούς που πραγματικά θα μπορούν να ωφελήσουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε όλες τις νέες περιφέρειες μάλλον σε όλε τι περιφέρειες και στι νέε περιφέρειες που θα έρθουν με την προσχώρηση τη Κροατία. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τι παρατηρήσει σα για τη συνεργασία. Προφανώ προσβλέπω να επιστρέψω στη δική σα την Επιτροπή και ελπίζω ότι θα έχω στα χέρια μου και μια έκθεση προόδου τότε, όταν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε του τριμερεί διαλόγου. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ κατανοούμε ότι το βλέπετε ξεκάθαρα ότι στο Ευρωκοινοβούλιο έχετε έναν εταίρο, ένα σύμμαχο που έχει τον ίδιο στόχο να μπορέσουμε να όχι να μόνο να, ολοκληρωθεί, να ολοκληρώσουμε το έργο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας αλλά από κοινού να πετύχουμε μια καλή δέσμη μέτρων για αυτή την πολιτική. Όχι μόνο από πλευρά κονδυλίων, αλλά και αυτό που καμιά φορά είναι πιο σημαντικό από ότι τα κονδύλια, να υπάρχει δηλαδή μια καλή θετική πολιτική που θα λειτουργήσει θετικά για την Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητά, ανταγωνιστικότητά της και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Προσβλέπουμε να σας ξαναδούμε περί τα τέλη της Προεδρίας σας μέχρι τότε ξανά οπωσδήποτε και ελπίζουμε θα έχετε καλά μαντάτα να μας δώσετε και που θα μπορούν να μας ικανοποιήσουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ελπίζουμε και σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχαριστούμε και για τον τρόπο με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις ε, διεξάγονται από τους συναδέλφους σας. Ευχαριστώ. Um, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τώρα και η δουλειά που έχουμε αφήσει, ένα σημείο το 7 που έχουμε αφήσει από την πρωινή μας συνεδρίαση. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Γιάν Όλμπριχ, το σχέδιο έκθεσής του για τη χορήγηση απαλλαγής για το 2011 όσον αφορά την ε, Επιτροπή. Έχεις τον λόγο Γιάν για να μας εξηγήσει τα σχετικά. Μάλιστα, ευχαριστώ. Όσοι ήθιστε σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε μέσα σε διαδικασία χορηγήση απαλλαγής που αφορά την Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε σχέση με εμά. Εμείς ως ε, Περιφερειακή Επιτροπή πρέπει να προετοιμάσουμε ως ήθιστε μια, ένα σχέδιο γνωμοδότησης με βάση την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Η γνωμοδότησή μας σύμφωνα με τους κανονισμούς είναι σχετικά σύντομη και αυτή η γνωμοδότηση βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα και στοιχεία από την ίδια την έκθεση που αντλούμε του ελεγκτικού συνεδρίου. Πολιτικά φυσικά υπό το πολιτικό πρίσμα υπάρχουν δύο τρόποι. Διτά μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί τα ίδια στατιστικά στοιχεία με δύο τρόπους. Οι συνάδελφοί μας από διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές που δεν είναι υπέρ της πολιτικής συνοχής θα χρησιμοποιήσουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία για να πούν ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ αρνητική, υπάρχουν τόσα πολλά σφάλματα κτλ. κτλ. Όλα αρνητικά λοιπόν. Εγώ στην γνωμοδότηση που προτείνω από πλευρά τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η πρόταση είναι απόλυτα σαφή. Στα σημεία αυτά έξι τα οποία εγώ προτείνω, είναι να πούμε ότι ακόμα και αν υπάρχουν κάποια σφάλματα ακόμη, θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ποια είναι τα αίτια αυτών των σφαλμάτων, να το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να διαφοροποιήσουμε αυτά τα πράγματα και προσπαθώ να υπογραμμίσω το πρόβλημα των παραβιάσεων όσον αφορά τους κανονισμούς και διατάξεις των δημόσιων προμηθειών πρόβλημα δηλαδή κρατών μελών στα κράτη μας. Επίσης να πούμε ότι είναι ένα σαφές προτέρημα αυτό. Η θετική αλλαγή, οι θετικές αλλαγές στην πολιτική συνοχή έναντι των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Αν δει κανεί την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, μπορεί να βρει τα αριθμητικά στοιχεία, τα δεδομένα που καταδεικνύουν ότι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερική Ανάπτυξης υπάρχει μια μεταβολή θετική μεταβολή όσον αφορά τα επίπεδα σφαλμάτων ή τα, το πιθανό επίπεδο σφάλματος. Γι' αυτό από πλευρά γνωμοδότησης ως πρώτο σημείο μπορείτε να δείτε ότι μειώνεται με φθήνουσα πορεία το στατιστικό σφάλμα. Και αυτό επίσης ε, είναι και αφορά και την ίδια τη μέθοδο όσον αφορά την ανάλυση. Στο σημείο 4 βρίσκεται την παρατήρηση που αφορά το πρόβλημα του επίπεδου σφάλματος που ε, χρησιμοποιείται και από το ελεγκτικό συνέδριο και φυσικά την προοπτική ε, που στο 2% και όχι θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους ελέγχους το ε, σύνηθες ε, επίπεδο ε, στατιστικού σφάλματος ήθισε να είναι 2%. Δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθεί αυτό. Το 2% λοιπόν που χρησιμοποιείται από το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθεί ο στόχος. Επίσης υπογραμμίζουμε και άλλα στοιχεία εδώ. Υπογραμμίζουμε τη μέθοδο που υιοθετεί, τις μεθόδους που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή του προγράμματος δράσης που είχε αποφασιστεί κατ' παρελθόν. Πρόκειται λοιπόν εδώ για το, α, την αύξηση του επίπεδου διακοπής και ε, παγώματος ε, ε, ακύρωσης και βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου ευπρόσδεκτο και έχουμε και την πρόταση να υιοθετηθούν ακόμα σκληρότερες μέθοδοι ώστε να υπάρξει αυτόματη διακοπή μετά από ε, εκπλήρωση κάποιων προϋποθέσεων. Τώρα συνεχίζονται αυτά και το τονίζουμε όμως θεωρεί το ελεγκτικό συνέδριο ότι η ε, πιστοποίηση ε, αξιοπιστίας ή ασφάλειας σε σχέση με το ποσοστό σφάλματος ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί αυτόματα να επιτευχθεί. Λοιπόν, γενικά τώρα υπό αυτό το πρίσμα αυτής της γνωμοδότησης υπάρχει μια σαφέστατη τάση να καταδείξουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες που καταβάλλονται, υπάρχουν οι θετικές τάσεις ε, που σημειώνονται, εξακολουθούν και υφίστανται προβλήματα όσον αφορά τις κρατικές δημόσιες προμήθειες από τα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν τα θετικά στοιχεία και έτσι καλοδεχόμαστε και ε, θεωρούμε ότι είναι ευπρόσδεκτες αυτές οι θετικές εξελίξεις. Αυτό το μήνυμά μας ως Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή άνθρωποι που είμαστε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως και οι θετικέ εξελίξεις και έτσι δεν αλλάζει η τοποθέτησή μας έναντι της ε, πολιτικής αυτής. Ε, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα ίδια στατιστικά στοιχεία θετικά και αρνητικά. Εμείς όμως είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι από πλευρά τη Επιτροπής ανάπτυξη γι' αυτό υιοθετούμε μια επικοδομητική στάση. Ευχαριστώ. Σκιώδης εισηγητές τώρα. Ο Αλφόνση πρώτο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι επί της ουσίας συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις του εισηγητού. Πράγματι. Είναι θετική δυναμική και αυτό είναι και το πρώτο που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχουν οι μηχανισμοί για έναν συστηματικότερο έλεγχο που είναι και μια σημαντική απέτηση ε, και των Ευρωπαίων πολιτών που θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται σωστά και γίνονται σεβαστοί οι στόχοι και οι διαδικασίες όμως. Γιατί αυτοί είναι οι δύο άξονες που μας απασχολούν. Θα ήθελα πάντως να πω στον εισηγητή, δεν ξέρω αν στα γαλλικά το κείμενο δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά στο σημείο 5 ε, ποιος είναι ο στόχος ακριβώς της παρατήρησης, δεν τον καταλαβαίνω να πάμε πιο μακριά, να αναλύσουμε περισσότερο, δηλαδή να επαληθεύσουμε ότι οι διορθωτικοί μηχανισμοί που αποφασίζονται από την Επιτροπή είναι δεδειγμένοι ή ότι πρέπει να τα θέσουμε όλα από αμφισβήτηση. Δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Η διατύπωση του σημείου 5 μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ίσως πρέπει να τη συζητήσουμε λίγο για να δούμε ακριβώς τι θέλουμε να πούμε με αυτό το σημείο 5. Κατά τα λοιπά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Μικάλη Τόιρερ. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ Ντανούτα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή Γιάνν Όλμπρεχτ για τη γνωμοδότηση αυτή. Υπό το πρίσμα της ομάδας Άλντε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στην ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου το ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται εξακολουθεί να είναι υψηλό και αυτό είναι ανησυχητικό στοιχείο. Όμως θετικά σημειώνουμε ότι μειώθηκε από το προηγούμενο επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε. Διότι οι διαρθρωτικές πολιτικές ε, πάντα ε, οι επικρίσεις ε, αφορούν τη μέτρηση αυτού του ποσοστού. Τώρα τα αίτια. Τα αίτια πρέπει να, επικεντρω... επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα αίτια ώστε να καταφέρουμε να μειωθεί, να μειωθεί τελικά αυτό το ποσοστό σφάλματος. Αυτό είπε και ο εισηγητής. 25% των, των πράξεων που ελέγχθηκαν κατέδειξαν σφάλματα. Όμως αυτό γίνεται μέσα στα εθνικά πλαίσια. Είναι υποχρεωμένο να σημειώνει αυτή την κατάσταση στο ελεγκτικό συνέδριο. Πρέπει ενισχυμένα η υπευθυνότητα των κρατών μελών να δράσει. Και βλέπουμε εδώ ότι για 80% των κονδυλίων που είναι σε αυτή την αρμοδιότητα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις και για την ε, ε, πληροφόρηση, ενημέρωση και το πρασίνισμα. Εμείς σε τριμερή διάλογο καταφέραμε να πετύχουμε τη δυνατότητα για την ε, απλούστευση, την διοικητική μπόρεσε να προχωρήσει. Και θα έπρεπε τώρα κοινό έργο μας να είναι, κοινό έργο όλων και στην τομεακή, στον τομεακό κανονισμό για τη διαθωτική πολιτική και τα διαθωτικά ταμεία αυτή η απλούστευση να μπορέσει να υλοποιηθεί συγκεκριμένα για τη χορήγηση απαλλαγής προς την Επιτροπή την οποία πρέπει να εξετάσουμε θα ήμουν ευγνώμων αν καταφέρναμε να πετύχουμε μια πλειοψηφία στο αίτημα ότι για το μέλλον πρέπει να έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο εμείς ως Κοινοβούλιο. Όχι μόνο να εξετάζουμε την νομιμότητα των πράξεων αλλά να εξετάζουμε αν η χρήση των κονδυλίων επιτυγχάνει το ευκταίο, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι νόμιμη και νομικά συμβατή η ε, δημιουργία ενός νέου αεροδρομίου. Αν όμως δημιουργηθεί ένα αεροδρόμιο και δεν προσγειώνονται αεροπλάνα και δεν υπάρχει κίνηση πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο, τότε είναι παράλογο, είναι χωρίς νόημα να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό η έκθεση λοιπόν σε σχέση με τα κονδύλια και την χρήση των κονδυλίων των διαθωτικών ταμείων κατέδειξε ότι σε κάποιο λιμάνι έγινε μία ε, προβλήτα, ή μία αποβάθρα που, χρησιμο... που χτίστηκε που δεν χρησιμοποιήθηκε όμως. Πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα τέτοιου είδους σφάλματα να μπορούν να επανορθωθούν ή να υπάρχουν κυρώσεις και πρόστιμα διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τέτοιου είδους λανθασμένες δράσεις να πολλαπλασιαστούν. Πιστεύω αυτά τα σημεία πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας στο έργο μας και προσπαθώντας να στραφούμε κατά των αρνητικών ε, παραδειγμάτων που αναφέρονται και αντίστροφα να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την βέλτιστη διαχείριση good governance και τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτές να επικεντρώνεται. Υπάρχουν πολύ περισσότερα θετικά τέτοια παραδείγματα και τότε εκείνοι που βρίσκονται ως ε, ε, το στο εδόλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική ας το πω προσέγγιση και προτού γίνει κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να οδηγηθούν στη λογοδότηση υπεύθυνη, διότι θα πρέπει εδώ να μπορέσει να ασκηθεί επιρροή στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες με αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κορνέλια Έρνστ στη συνέχεια παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ καταρχήν. Πρώτα προς τον ίδιο τον συντάκτη γνωμοδότησης για αυτό το φλέγον θέμα Λοιπόν, γίνεται λόγος για μεγάλο σφάλμα, στατιστικό σφάλμα και πρέπει να υπάρξουν περικοπές στα κονδύλια της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη και τη συνοχή. Είναι πολύ δύσκολο και ακαθόδε αυτό το θέμα. Όταν αναφέρεται ότι τα αίτια του ποσοστού σφάλματος πρέπει να αποσαφινιστούν και να καταδειχθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό είναι λόγος ύπαρξης για μας είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Το δέχομαι αυτό, με κάποια πράγματα, πράγματα έχω κάποια προβλήματα. Αφορά το σημείο 5 αυτή η παρατήρηση το να σταματήσουν ή να, παγωθούν, ε, να παγώσουν οι πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σημειώνουμε αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να δούμε είναι η σωστή πορεία αυτή έτσι να αντιδρούμε μια τέτοια πολιτική να υιοθετούμε. Στο σημείο 5 θα ήθελα να πείτε δύο λόγια. Πολυσχηδώ υπάρχουν ασάφειες. Ένα συνάδελφος είπε πώς θα υπάρχει αντιστάθμιση η εύλογη, η ε, θεμητή αντιστάθμιση. Πώς θα μπορούν τέτοιου είδου φάλματα να αντισταθμιστούν. Δεν θα μπορούσαμε να εγγυηθούμε ότι κτλ. Εδώ υπάρχει ασάφεια. Και για το τελευταίο σημείο το απορρίπτω, για τον εξή λόγο. Χαιρετίζω όλε τι προσπάθειε βέβαια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει ενίσχυση τη απλούστευση. Αλλά εξ άντε τώρα, σε σχέση με την, την πιστοποίηση και όλα αυτά τα οποία συναρτώνται με τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες να υπάρξουν ε, περικοπές ε, το αν αυτό συνεισφέρει για απλούστευση αμφιβάλλω πραγματικά. Και εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε στο συνολικό πρόβλημα για την πολιτική συνοχή. Να δούμε με συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία από πλευρά κρατών μελών θα πρέπει να ε, υποβάλλονται. Δεν δημιουργούμε εμείς μια πηγή σφάλματος με αυτόν τον τρόπο και έτσι μετά είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν σφάλματα. Ευχαριστώ. Mm. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και διαρωτώ με, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να παρέμβει επίσης. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Αλλά προτού παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 168 του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου και το 160, τι είναι το ποσοστό των συνολικών πληρωμών, τι, ποιο ποσοστό συνολικών πληρωμών είναι αυτό, μπορείτε να μας πείτε, έχετε τον λόγο τώρα γενικά για τα σχόλιά σας, για τα θέματα που συζητούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστήσω και τον κύριο Ολμπρίχτ για το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την απαλλαγή. Είναι πολλά τα ενδιαφέροντα στοιχεία της γνωμοδότησης και σας ευχαριστούμε και για την υποστήριξή σας βέβαια. Η πολιτική συνοχής τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε αντικείμενο έντονη κριτική σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δημοσιονομική διαχείριση, δικαιολογημένα ενίοτε και κάναμε τεράστιε προσπάθειε, το αναφέρατε, μετά το σχέδιο δράση του 2008, τόσο ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το ποσοστό σφάλματος συνολικά για τη συνοχή είναι στο κεφάλαιο 1 φέτος στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο έχει κάνει μια διάκριση για το ΦΕΝΤΕΡ, Ταμείο Συνοχής Κοινωνικό Ταμείο, στα διάφορα ταμεία το έχει ε, υποδιαιρέσει. Έχουμε ένα ποσοστό εδώ για να κάνουμε μια σύγκριση με το προηγούμενο έτος για το most likely error, το πιο πιθανό σφάλμα, 5,1% σε σύγκριση με 7,7% κατά το περσινό έτος. Άρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Στο κεφάλαιο 6 για το κοινωνικό ταμείο και για το ΦΕΝΤΕΡ. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό το ΕΤΠΑ δηλαδή, που δεν κρύβεται πίσω από τη βελτίωση του έκτα, Βλέπουμε βελτίωση συνολική για όλα τα ταμεία. Επίσης, ήθελα να σας ε, αναφέρω ότι στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΤΖΟ υπολογίζει τον κίνδυνο μεταξύ του 3,1 ε, και του 6,8 για το 2011. Αυτή είναι η ψαλίδα του ποσοστού σφάλματος ε, που μας μετέφερε το ελληνικό συνέδριο. Και αυτό πρέπει να το συγκρίνουμε με, ένα, μια οροφή για το 2006-2008 ε, της τάξης του 11% που ήταν και το ποσοστό ε, το κατώτερο ποσοστό σφάλματος. Τεράστια βελτίωση δηλαδή. Βελτίωση που λέει και ο κύριος Όλμπριχτ στην έκθεσή του ότι σχετίζεται με συγκεκριμένα στοιχεία και πρώτα απ' όλα πολύ πιο αυστηρή πολιτική εποπτείας από τη ΓΔ και βλέπουμε πια ότι και τα νομικά μέσα χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται άπαξ και ε, διαπιστώσουμε προβλήματα. Το 2012 η ΓΔ έχει μπλοκάρει και πληρωμές ε, σε 190 προγράμματα και έχει και 156 ε, διαδικασίες. Ε, για δύο ε, προχώρησε σε αναστολή. Επομένως προχωρούμε και έχουμε και το σχέδιο δράσης με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που εντοπίζουμε. Και η αναστολή των πληρωμών σταματά μόνο όταν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για το ότι διορθώθηκε το πρόβλημα. Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλές άλλες δράσεις, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρω και κάτι ακόμη. Το εύρος δηλαδή των προβλημάτων, διότι στο σχέδιο ψηφίσματος ε, μιλάτε για συχνότητα ε, σφαλμάτων. Πρέπει να σας πω ότι το ελεγκτικό συνεδρίο έχει ένα δεύτερο δίκτυ ε, που είναι συχνότητα των σφαλμάτων 59%, 59 για το ΕΤΠΑΛΑ πιάνει όλα τα σφάλματα, από το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σοβαρό, από αυτό που έχει σχεδόν μηδενικό οικονομικό αντίκτυπο μέχρι αυτό που έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο που καθιστά μη επιλέξιμο ένα σχέδιο. Και θα πρέπει αυτό το δίκτυ να τον εξετάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή. 59% λοιπόν των σχεδίων από τα 168 ε, βλέπαμε ότι είχαν τουλάχιστον ένα σφάλμα που μπορεί να ήταν απλά μια καθυστέρηση στη δημοσίευση μιας προκήρυξης διαγωνισμού. Προβλέπονται 45 ημέρες στον κανονισμό. Αν ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τρεις μέρες μετά, αυτό θεωρείται τυπικό σφάλμα και καταμετράται. Αλλά δεν επηρεάζει καθόλου τον προπολογισμό ή την ε, ορθή υλοποίησή του. Βέβαια έχουμε και ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, που και αυτά λαμβάνονται βέβαια υπόψη. Και σε ό,τι αφορά αυτά ποσοτικοποιήσιμα, τα ποσοτικώ μετρήσιμα σφάλματα, τα σχέδια τα οποία αποβάλλονται σε νησμούς και που βλέπουμε να παρουσιάζουν τέτοια σφάλματα είναι πάνω από το 50% των σφαλμάτων για το ΕΤΠΑ. Πάνω από το 50% δηλαδή του 5,1 προέρχεται από προβλήματα που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις που δεν εφαρμόζονται δηλαδή σωστά από τα κράτη-μέλη. Τελευταίο σημείο που είναι σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε το 62% των σφαλμάτων για το ΕΤΠΑΘ λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί με επαλήθευση σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτο βαθμό. Και πρέπει να υπενθυμίσω στους βουλευτές ότι εκτιμά το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξάντε προποθέσει και θα σα πω και κάτι ακόμη. Οι επαληθεύσει, οι έλεγχοι των διαχειριστικών αρχών εξάντε δηλαδή, είναι προπόθεση εκ των όνων κάνευ για να μειωθούν τα σφάλματα. Γι' αυτό και συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε. Το 62% των σφάλμα θα μπορούσε να μειωθεί με τις επαληθεύσεις, αν γίνονταν επαληθεύσεις ε, σωστά και αν ήταν αποτελεσματικές. Για το σημείο 5 τώρα, η φράση που αναφέρεται προέρχεται από την έκθεση 3 του 2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκανε λόγο για την δυνατότητα της Κομισιόν να διορθώσει, για τη διόρθωση. Είχαμε δει ε, το 2006 πάνω, ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Είχε εντοπίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτά τα προβλήματα και η Κομισιόν προέβη σε οικονομικές διορθώσεις και τροποποίηση των προγραμμάτων. Όμως το συνέδριο θεώρησε πολύ νωρίς για το κλείσιμο του 2006 για να δούμε κατά πόσον οι οικονομικές διορθώσεις αντιστάθμιζαν επαρκώς τον κίνδυνο που είχαν εντοπίσει στη συγκεκριμένη περίοδο. Υποσχεθήκαμε λοιπόν ε, στον εισηγητή και στην Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού να δημοσιεύσουμε μία έκθεση για το ποσοστό σφάλματος για τη χρήση για το 2006 και για το ε, για τις διορθώσεις που κάναμε και να δούμε πώς επηρέασαν οι διορθώσεις αυτές τα προγράμματα. Δεύτερη πτυχή. Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθούν να υπάρχουν προγράμματα που τακτικά ε, δημιουργούν προβλήματα, εμφανίζουν προβλήματα. Ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε αυτή τη διαπίστωση, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δούμε το ποτήρι και μισογεμάτο αλλά και μισοάδιο. Το μισογεμάτο ποτήρι λέει ότι υπάρχει βελτίωση, έχουμε μείωση του ποσοστού σφάλματος στην περίοδο 2007-2013 και αυτό είναι μια απόδειξη. Μια βουλευτής ε, που μίλησε πριν από τη Σαξονία ε, πρέπει να πω ότι για το πρόγραμμα αυτό το 94-95 είχαμε τεράστια προβλήματα οικονομικά και με το κρατήδιο αυτό της Αξονίας ε, συνεργαστήκαμε και γι' αυτό σήμερα το πρόγραμμα της Αξονίας είναι εξαιρετικό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να διορθώσουμε τα προγράμματα, να αναφέρουμε και την Ελλάδα που όπως θα δείτε στην έκθεση ε, υπέστη σημαντικές δημοσιονομικές διορθώσεις ε, από το 2000 στο 2006 αλλά και το ίδιο βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση δηλαδή το 2007-2013. Όπου υπάρχουν προβλήματα έχουμε συχνά έλεγχο, λογιστικό έλεγχο και επικεντρωνόμαστε βέβαια στους κινδύνους για να διορθώσουμε τα πράγματα. Το ποσοστό του 2011 δεν μας δείχνει να έχουμε συγκέντρωση σφαλμάτων σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Αντίθετα με αυτό που είχαμε πει σε ένα κείμενο ανάλυσης πέρυσι για τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό διότι οι διορθωτικές μας δράσεις, διακοπές, αναστολές μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη βάση του, στη ρίζα του. Προτού υπάρξει δήλωση και επιληφθεί το, το ελεκτικό. Δεν μπορεί να επιλέξει δηλαδή το ελεκτικό συνέδριο αυτές τις ε, σφαλμένες πληρωμές. Όλες αυτές οι δράσεις λοιπόν πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε ε, τον εισηγητή για το σχέδιο ψηφίσματος που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό. Και θέλω να σας πω ότι στο Συμβούλιο, όπου συζητούμε επίση το σχέδιο ψηφίσματος ε, του Συμβουλίου, λέει ο μιλητής, υπάρχει πάλι αυτή η διχοτόμηση. Κάποια κράτη-μέλη βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, κάποια το βλέπουν μισοάδιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Όλμπριχτ που ε, τάχθη υπέρ ε, της πολιτικής μας ε, και που θα μας βοηθήσει και στο μέλλον και να επικεντρώσουμε το αποτέλεσμα στην αποτελεσματικότητα, στην αποδοτικότητα, αφού βέβαια ενισχύσουμε το σύστημα και λύσουμε το πρόβλημα με την ε, κανονικότητα και την νομιμότητα, που ακόμα δεν το έχουμε λύσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν έχει τελειώσει η συζήτηση γιατί βλέπω ότι ενέπνευσε η παρουσίαση του εκπροσώπου της Κομισιόν και άλλους ομιλητές ε, ο κύριος ε, Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα. Χαιρετίζω, χαιρετίζω την έκθεση του κύριου Όλμπρεχτ. Κάποιες παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Εκκινώντας από το τέλος αυτής της ε, γνωμοδότησης, πώς διαπιστώνετε πώς διαμορφώνεται η απεικόνηση της πραγματικής κατάστασης ε, με μια μείωση που θέλουμε να πετύχουμε του ποσοστού σφάλματος. Υπάρχει όμως ίσως ε, και κάποια υπόνοια καταχρήσεων ή ε, καταχρήσεων κονδυλίων ή τι θα γίνει σε σχέση με ε, δραματικές διαστάσεις που μπορεί να, δίνεται, να δίνονται σε σφάλμα, σε ποσοστό σφάλματος που θα ξεπερνά το μηδενικό ποσοστό. Εμείς ε, ως πολιτικοί πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα. Υπάρχει η ανάγκη, το δυναμικό, το διοικητικό και ε, δυναμικό ε, δράσης ε, του επίπεδου ενός προγράμματος πρέπει να μπορεί να αναβαθμίζεται. Όμως ε, όταν υπάρχουν τέτοιες ελπίδες η ελπίδα πεθαίνει τελευταία πάντα, όταν έρθει η ώρα της όμως πεθαίνει. Όταν έχουμε τη νέα περίοδο προγράμματος, προγραμματισμού μετά το 2014 σε κάθε κανονισμό για κάθε ταμείο θα πρέπει να εμπεριέχεται κάτι για την αύξηση του διοικητικού και διαχειριστικού δυναμικού και πρέπει να δούμε και κάποιες από τις περιπτώσεις κατά τα άλλα στις οποίες ε, ε, υπήρξαν προβλήματα για παράδειγμα όσον αφορά και το μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε να αντιδράσουν οι αρχές κάποιου κράτους μέλους ε, π.χ. έστω από τη Ρουμανία ή για συστάσεις ε, ή προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι πρέπει να γίνει σε σχέση με τη δυνατότητα αντίδρασης από τις κρατικές αρχές. Αυτά πρέπει να συνδεθούν με τα θέματα διαχείρισης ε, και ελέγχου είτε από πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο είτε από άλλη διοικητική αρχή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η πτυχή σε σχέση με ε, έγγραφα τα οποία αφορούν τέτοιου είδους δράσεις από το καλοκαίρι του 2011 και μόνο το φθινόπωρο ε, υπευλήθη απάντηση και διέτρεξε κινδύνους να απολέσει τα κονδύλια συνοχής ε, η Ρουμανία. Δεν έγινε τίποτα όμως το 2010. Υπήρξε μια πολύ αποδυναμωμένη αντίδραση και ικανοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με κάποιες συζητήσεις κάποιες φήμες που κυκλοφορούσαν. Πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαζώσεις να πει ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει, πότε πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αντίδραση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέτοιες καθυστερήσεις πρέπει να είναι άμεση και ε, κάθετη και θα έπρεπε να οδηγεί σε απόφαση να παγώνει ή να ε, πάβει η χορήγηση τέτοιων κονδυλίων. Αλλά ποιος θα πληρώσει. Η κοινότητα θα πληρώσει στο τέλος τέλος αν όλα αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο, στην απορροφητικότητα και την ικανότητα απορρόφησης ε, κονδυλίων από πλευράς μιας χώρας. Πιθανότατα η ικανότητα απορρόφησης ε, μπορεί να πλησιάζει μηδενικό ποσοστό σε τέτοιου είδους περιπτώσεις προβλημάτων. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη τελικά να αντιδρούν σε τέτοιου είδους προειδοποιήσεις και κρούση κόδωνα κινδύνου. Και επίσης ε, μια αντίδραση σε σχέση με τις πελατειακές σχέσεις που μπορεί να υφίστανται. Αυτό βαίνει εκ παραλίλου με υπόνοιες ε, για κάποιες απάτες. Πολλές φορές ε, υπάρχει κάποιος νεποτισμός, υπάρχει τέτοιου είδους ευνοιοκρατία. Δεν συμβαίνει αυτό μόνο στην Ρουμανία, συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες σε σχέση με κανονισμούς εθνικούς ή εταιρείε που εμπλέκονται ε, σε σχέση για παράδειγμα με τα όσα τεκταίνονται είτε στη Ρουμανία είτε αλλού. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να καθορίσουμε επακριβώς ε, πώς θα πρέπει να αντιδρούμε σε τέτοιου είδους ε, καταστάσεις όσον αφορά εργολαβίες και υπεργολαβίες και σε σχέση με τα προϊόντα παραγωγή αγαθών αλλά και με την παροχή υπηρεσιών. Υπάρχουν απάτες πολλές φορές επειδή οι μονάδες αντιμετώπισης της κρίσης θα πρέπει άμεσα να δρούν όταν υπάρχει κάποια τέτοια υπόνοια ή κάποια στοιχεία για τέτοιου είδους απάτες ή παρατυπίες. Αυτό θέλουμε να γίνεται με προσόφερος του κοινού στόχου. Να υπάρχει ένα υγιές ποσοστό απορρόφησης και να μειωθεί το ποσοστό απατών και παρατυπιών. Και θέλουμε πάνω απ' όλα, κύρια και πρότιστα, να βελτιώσουμε το ποσοστό απορρόφησης, απορροφητικότητας, όπως είπε και ο Γιάννη Όλμπριχτ. Ποσοστό απορροφησης των των ε, Ευρωπαϊκών Ταμείων. Δεν θέλουμε να συμβαίνει το οτιδήποτε, αλλά αυτό συγκεκριμένα να μπορέσουμε να επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στη συνέχεια, μετά από όλα αυτά που αναφέρθηκαν και από πλευράς ε, Τόιρερ και Μποστινάρου, και σε σχέση με αυτά τα οποία μας παρουσίασε ο κύριος Γιάνν Όλμπριχτ. Πρέπει να προσέξουμε θα έλεγα εμείς την πολιτική συνοχή και την διαθοτική πολιτική να μην την υποβαθμίσουμε ή να μην δεχθούμε να ε, βρεθεί υπό υπόνοιες. Ε, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η διαθοτική πολιτική και η πολιτική συνοχή ιδιαίτερα για τις περιφέρειες που απειλούνται από την κρίση ή ε, υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και πρέπει εκεί να παρεμβαίνουμε. Ωστόσο όμως αν διαβάζει κανείς κάποια δημοσιεύματα πως για παράδειγμα από τις τους ελέγχους του ελεγκτικού συνεδρίου μέγιστος αριθμός ε, ε, καλύπτεται από ε, υπερβολικά σφάλματα και μετά κραυγάζουν ότι υπάρχει διασπάθηση κονδυλίων πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να δούμε όπου υπάρχουν καταχρήσεις, όπου χρήματα χρησιμοποιούνται για παράλογα σχέδια, ε, πρέπει να δρούμε και δεν επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο και να δεν πρέπει να το επιτρέπουμε και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με ποσοστά σφάλματος. Ο συνάδελφος Σόλμπριχτ είπε πολλές φορές αυτά συναρτώνται με το δίκαιο, εθνικό δίκαιο των κρατών μελών όσον αφορά κρατικές προμήθειες και συμβάσεις. Έχουμε ένα εμβαλωματικό τοπίο ενώπιόν μας που συναπαρτίζεται από 27 κράτη-μέλη. Από δικές μου σκέψεις και προβληματισμούς γνωρίζω πώς ε, συνεργάτες επιτόπου στα κράτη-μέλη εκφοβίζονται και τους λένε αν γίνει κάποιο λάθος, κάποιο σφάλμα και είναι υπάλληλοι αυτοί μπορεί να απαιτηθεί η ανάκτηση κονδυλίων, η επιστροφή κονδυλίων και εσείς οι ίδιοι υπάλληλοι θα είσαστε υπεύθυνοι για κάτι τέτοιο και τότε λένε οι υπάλληλοι α δεν θέλω τότε να έχω καμιά σχέση με ένα τέτοιο θέμα. Η πρόβλημα. Πρέπει να αποσοβήσουμε ένα τέτοιο κίνδυνο και να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά σε αυτό το κομβικό σημείο. Ήρθε η χρονική στιγμή, νομίζω, προπαρασκευάζοντας την μελλοντική πολιτική μας, να εναρμονίσουμε το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις και τις κρατικές προμήθειες στην Ευρώπη. Διότι αυτό μου φαίνεται να είναι το σημαντικότερο στοιχείο αυτή τη στιγμή. Εκεί διαπιστώνονται ε, περιπτώσεις σφαλμάτων που είναι υπερβολικά και που μπορεί αυτό να οδηγήσει η εμπλοκή και ο ζήλος των χαμηλότερα στην ιεραρχία των χαμηλότερων υπαλλήλων να απειληθεί η δράση τους ε, ή να φοβηθούν και να μην δράσουν όπως πρέπει. Ένα άλλο θέμα είναι η ελεγκτική δράση των ελεγκτών. Λέμε σαν να είναι το ελεγκτικό συνέδριο ένα ε, θεϊκό όργανο, ένα είδους ας το πω έτσι ε, όργανο που είναι, ό,τι λέει είναι θέσφατο. Πρέπει αυτό να το επανεξετάσουμε. Στις γενικές διευθύνσεις θα πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα και ανοιχτό πνεύμα ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε, αλλά δεν κατάλαβα με καταλάβατε καλά όταν προηγούμενα διατύπωσα την ερώτησή μου. Θα ήθελα να ξαναδιατυπώσω αναδιατυπώσω την ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μία δέσμη προγραμμάτων, σχεδίων ή πληρωμών επιλέγεται από το ελεγκτικό συνέδριο για τέτοιου είδους ελεγκτική χρήση, υπάρχει μία τέλεια ιδανική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το ελεγκτικό συνέδριο και δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Παρόλα αυτά όμως τούτων λεχθέντων θα ήθελα να κατανοήσω καλύτερα ποιο ποσοστό είναι αυτό του συνολικού αριθμού πληρωμών αν αναφερθούμε σε ένα τέτοιο έτος ελέγχου ποιο ποσοστό για παράδειγμα του 2011 των πληρωμών διαπιστώνεται ότι από το ε, δείγμα αυτό που εξετάστηκε δειγματοληπτικά από το ε, ελεγκτικό συνέδριο 168 για παράδειγμα πληρωμές που κατά το έτος αυτό επελέγησαν προς έλεγχο. Ποιο ποσοστό αυτών των πληρωμών του συνολικού αριθμού πληρωμών είναι εκείνο το οποίο ελέγχθηκε σε σχέση με αυτόν τον αριθμό των 168 πληρωμών. Μπορείτε να μου δώσετε αυτό το στοιχείο στην απάντησή σας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Νόμιζα ότι αναφερόσταν στη συχνότητα. Ε. Όχι, και αυτά που μας είπατε ήταν πολύ ενδιαφέροντα, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχω τον αριθμό των πληρωμών που έκανε η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Μιλάμε πάντως για χιλιάδες ε, πληρωμές για όλα αυτά τα προγράμματα του ε, Ταμείου συνοχή καθώ επίση και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξη, τα οποία ελέγχει το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο όμω ασχολείται και με άλλα ταμεία. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση θα μπορούσε να σας δώσει το ελεκτικό συνέδριο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι χρησιμοποιεί περίπου ένα δείγμα 180 συναλλαγών που θεωρούνται τελικά αρκετά αντιπροσωπευτικέ για όλο το φάσμα των πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποφανθεί για τη μεθοδολογία του ελεκτικού συνεδρίου. Η μεθοδολογία πάντω αυτή χαρακτηρίζεται ω αποδεκτή μέθοδο όσον αφορά τα πρότυπα ελέγχου. Μία παρατήρηση μόνο μπορώ να κάνω. Όπω ξέρετε, οι ελεκτικέ αρχέ των κρατών μελών χρησιμοποιούν επίση στατιστικά δείγματα για ομάδε προγραμμάτων. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τα στατιστικά δεδομένα είναι να έχουμε δείγματα ομοιογενή προκειμένου να μπορούμε να καταλήγουμε σε σωστά συμπεράσματα. Βέβαια, όταν κάνετε έλεγχο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις πληρωμές προκύπτουν κάποια προβλήματα. Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε σωστά όλα τα σφάλματα. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα ένα λάθος το οποίο θα, θα μπορούσε να αντιστοιχίσει σε ένα ποσοστό σφάλματος 100% δεν σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να είναι επιλέξιμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σφάλμα το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% του συνόλου των προγραμμάτων για την Ευρώπη. Όταν σας λέω λοιπόν ότι οι δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούν σε πάνω από το ίμιση του ποσοστού σφάλματος, ουσιαστικά αναφέρομαι εδώ πέρα σε προγράμματα τα οποία μπορεί να έχουν παρουσιάσει σφάλμα της τάξης ε, σε υψηλότερο ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιλέξιμα τα προγράμματα αυτά, αλλά ότι μπορεί να έχει προκύψει ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού. Ακολουθούνται πάντως εδώ πέρα από το λεκτικό συνέδριο και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Πρόεδρος, Δηλαδή για τα περισσότερα από τα 300 προγράμματα στα πλαίσια του ERDF θα πρέπει κάθε φορά να έχουμε εκατοντάδες προγράμματα προκειμένου να γίνει σωστά ο έλεγχο. Ενδεχομένω, ουσιαστικά εδώ πέρα να αναφερόμαστε σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Αν πούμε ότι το σύνολο των προγραμμάτων τελικά μπορεί να φτάνει ακόμα και τα χίλια, να ξεπερνά τον αριθμό αυτό. Ο Γιάννη Όλμπριχτ θέλει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσπαθούσα και εγώ να βρω κάποια αριθμητικά δεδομένα στην έκθεση έχουμε έναν αριθμό πληρωνών 32.000 για την περιφερειακή πολιτική και περίπου 1.000 όσον αφορά την πολιτική μεταφορών, 900 για την ενέργεια, σε σύνολο χιλίων το δείγμα είναι 180. Αυτή λοιπόν είναι η μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί. Εμείς ε, πέρα από πολιτική Θέλουμε να πιστεύουμε όλα στη μέθοδο αυτή ότι είναι όντως μία μέθοδος αντι, αντικειμενική και αντιπροσωπευτική. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι κάποια κράτη-μέλη βρίσκονται πιο συχνά στο δείγμα από κάποια άλλα. Αυτό δεχομένως να συμβαίνει τυχαία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας πάντως και θα ήθελα πολύ γρήγορα να απαντήσω σε κάποια πράγματα. Πρώτον, η συνήθις διαδικασία είναι ότι Ακούμε το ελεκτικό συνέδριο, καθώς επίσης και τα όσα έχει να πει η Επιτροπή Προπολογισμών, ελέγχου του προπολογισμού. Δεν μας ενδιαφέρει όμως εδώ πέρα μόνο το επίπεδο του σφάλματος, η μεθοδολογία, αλλά και το πώς μπορούμε να καταμετρήσουμε την, την αποτελεσματικότητα και πώς μπορούμε να καταλήξουμε τελικά σε προγράμματα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά και θα έχουν χαμηλά επίπεδα σφάλματος. Νομίζω ότι ε, δεν μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή μία μαγική λύση, ούτε το λεκτικό συνέδριο μπορεί να μας δώσει αυτή τη στιγμή μια μοναδική απάνταση. Από ό,τι φαίνεται πάντως και το λεκτικό συνέδριο εστιάζεται όχι μόνο στο επίπεδο σφάλματος αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για απάτη. Με την απάτη ασχολείται Όλαφ. Το ελεκτικό συνέδριο ασχολείται με το σφάλμα. Σφάλματα και απάτη δεν είναι το ίδιο πράγμα, α μην τα συγχαίουμε και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Διαφορετικά καταλαβαίνω ότι καταλήγουμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν δείτε την πρόταση γνωμοδότησή μου, θα δείτε ότι καταρχά αναφέρομαι στο ζήτημα τη συχνότητα, πάνω από 50%. Στη συνέχεια όμω λέμε τι θα πρέπει να γίνει στην τελική αξιολόγηση, γιατί και η συχνότητα από την, από την άλλη δεν είναι ιδιαίτερα την προσωπευτική ω προ την πραγματική κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο άκουσα και πολύ προσεκτικά τις παρατηρήσεις σας για το σημείο 5. Όντως η διατύπωση εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολύ σαφής. Λέμε ότι γίνεται μια θετική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το Λοπτικό Συνέδριο από τη δική του πλευρά πιστεύει ότι δεν αντισταθμίζονται παρκώς τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί και το καθεξής. Νομίζω ότι πρέπει, ε, αν πάτε μάλλον στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, θα ακούσετε εκεί ότι οι συνάδελφοι ζητάνε όλο και περισσότερες διορθώσεις, περισσότερους ελέγχους, λιγότερα χρήματα για τη δική μας την πολιτική, όλο και περισσότερες αναστολές και διακοπές των πληρωμών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε επιτέλους αυτό το σχέδιο δράσης, το οποίο τελικά θα είναι αποτελεσματικό και θα διορθώσει αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Θα τώρα για την τελική εκδοχή του σχεδίου αυτογνωμοδότησης. Το σημαντικό είναι να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Σαφώ υπάρχουν εσφάλματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν, αλλά δεν θα πρέπει να αλλάξει γενικότερη στάση για την πολιτική μα. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να αποφασίσουμε και για την ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών. Εγώ σας προτείνω την 28η Ιανουαρίου. Δεν ξέρω ποια μέρα είναι, μάλλον Δευτέρα. Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Αυτή λοιπόν η καταλεκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης συζήτηση με τον συζητητές για τις κοινέ διατάξεις για τα ευρωπαϊκά ταμεία που ξέρετε ότι αυτός είναι ο γενικός μας λεγόμενος κανονισμός Έχουμε δώσει σε όλα τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη της, Ευρωπαϊ... της Επιτροπής μας τον πίνακα αυτό με τις τέσσερις στήλες, όπου βλέπετε το κείμενο που αντιστοιχεί στην έκβαση των διαπραγματεύσεων, καθώς επίσης ε, και τους ε, προσωρινούς συμβιβασμούς για διάφορα ζητήματα. Και ελπίζω ότι αυτό θα διευκολύνει τα πράγματα για τον Λάμπερτ Βανίστερόι, που είναι ο εισηγητής μας, ο οποίος θα μας ε, παρουσιάσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η Κωνσταντσα δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί στη σημερινή συζήτηση, επομένως είναι ο Λάμπερτ αυτός ο οποίος θα μιλήσει και εξ ονόματός της. Λάμπερτ, έχει το λόγο και μετά τη δική σου παρουσίαση νομίζω ότι θα έχουμε και λίγο χρόνο για να κάνουμε και κάποια συζήτηση. Πρέπει στις 6 ώρα πάντως να ολοκληρώσουμε γιατί ακολουθεί μετά και η συνεδρίαση των συντονιστών. Αν δεν μας μείνει πολύς χρόνο σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και αύριο. Λάμπερτ Βανίστερόι. Σας ευχαριστώ. πολύ. Αυτή τη χρονική στιγμή μπορούμε ακριβώς ε, με ακρίβεια να αναφέρουμε αυτό το οποίο συμφωνήθηκε κατά τα τέλη του 2012 και υπό την Κυπριακή Προεδρία. Και καθώς έχουμε συμφωνήσει με βάση την εντολή να εργαστούμε, είναι απόλυτα σαφές. Πήραμε αυτή την εντολή ακριβώς ως είχε και διαπραγματευθήκαμε με βάση αυτή την εντολή και στη συνέχεια αυτό μας δίνει αυτή τη θέση. Όλα τα κείμενα που παρουσιάζονται και όλα τα μέλη, όλοι οι ευρωβουλευτές και οι κοινοβουλευτικές ομάδες που έχουμε αυτή την έκβαση ενώπιόν μας, αυτά είχαν συμφωνηθεί σε ένα, ε, ένα βράδυ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων αργά το βράδυ για αυτό το θεματικό πλέγμα για το στρατηγικό προγραμματισμό και σχεδιασμό με την συνένεση από την άλλη πλευρά των σκιωδών εισηγητών που ήταν παρόντες. Και τώρα ίσως, όχι τώρα για να επαναλάβουμε αρχές από αυτών, είναι όμως ε, λογικό και συνετό να, αναφερθεί κανείς σε αυτά τα άρθρα εξειδικευμένα και να δει κανείς τι γίνεται σε σχέση με τα κείμενα και την ε, προοπτική για συμβιβασμό. Γιατί αυτό είναι ακριβώς το έργο που πρέπει να επιτυγχάνεται σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Ας αναφέρω σύντομα λοιπόν αυτά τα άρθρα ένα προς ένα και ας περάσω μετά στο ότι Αυτά τα στοιχεία, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να ενταχθούν στη συζήτηση και θα είναι πιο εύκολο σε υστερότερη φάση να μπορέσουμε όλα αυτά να τα εντάξουμε όπως ευελπιστώ στην επόμενη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί όταν θα έχουμε ολοκληρώσει με τα άλλα τμήματα τα οποία βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση. Άρθρο 1. Λοιπόν, ήδη το όνομα εδώ, ο τίτλος ε, και ε, η επίτευξη συμφωνίας επ' αυτού ευρωπαϊκά ταμεία, διαθροτικά ευρωπαϊκά ταμεία και επενδυτικά ταμεία. Ακούσατε τη νέα Προεδρία την Ιρλανδία δηλαδή υπό αυτό το ίδιο πνεύμα να τοποθετείτε. Τώρα η δική μας ιδέα η δική μας ιδέα είναι αυτά τα επενδυτικά ταμεία, αυτές οι επενδύσεις να μπορέσουν να, ε, να γεφυροποιήσουν σε σχέση με αυτά τα στοιχεία της ανάγκες. Εξετάζουμε αμφίδρομα τους ορισμούς και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι και στην μακρο, μακροοικονομική στρατηγική και στην περιφερειακή στρατηγική τα κείμενα αυτά ήταν, στοχεύαμε να είναι η βάση ενός συμβιβασμού και έπρεπε να εξεταστούν και κάποια άλλα σημεία και κατέληξε το Συμβούλιο με κάποιες ιδέες που παρουσίασε για συγκεκριμένες συστάσεις και συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, το άρθρο 2, καθώς ε, εμείς πιστεύουμε, είναι απόλυτα αποδεκτός έχει τώρα. Το άρθρο 4, πολύ σημαντικό για την θέση της εταιρική σχέσης, πώς θα λειτουργεί η εταιρική σχέση. Σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο είπε ναι εντάξει όμως πρέπει να σεβαστείτε από πλευρά σας το θεσμικό νομικό πλαίσιο σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Απόλυτα ορθό αυτό. Υπάρχουν κράτη που εργάζονται με ένα εθνικό πρόγραμμα και υπάρχει τελείως διαφορετική δομή για παράδειγμα σε ένα ομοσπονδιακό κράτος επ' αυτών. Αυτό που διατηρήσαμε λοιπόν τελικά ποιο ήταν. Αυτό που θεωρούσαμε εμεί σημαντικό για την εταιρική σχέση, για τους εταίρους μας, σε σχέση με τα αιρετά σώματα, όσον αφορά για παράδειγμα πόλεις, ε, δήμους, κοινότητες και όσον αφορά τα θέματα της εδαφικής συνοχής ε, και της περιφερειακής συνοχής Τώρα, η αρχή της επικουρικότητας που διαρκώς αναφερόταν ως θέμα από πλευράς ε, της, του Συμβουλίου και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο εκ με τα εθνικά προγράμματα αναθεώρησης ε, και στο άρθρο 5 πάλι τι έχουμε μπροστά μας. Πάλι ε, η εταιρική σχέση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η διαχείριση και σε σχέση με τη συζήτηση ένα κείμενο το οποίο θα σέβεται τους εθνικούς κανονισμούς και διατάξεις ως έχει η πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατηρήσαμε τις κυριότερες αρχές μας στο κείμενο και έχουμε και συμφωνία σε σχέση με τους εταίρους που είναι πιο σημαντικοί για τους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις αυτού του σχεδιασμού και της προπαρασκευής για την υλοποίηση των στόχων της περιφερειακής πολιτικών αυτών στην περιφερειακή πολιτική. Και στο άρθρο 5 αναφορά στο δεοντολογικό κώδικα. Πραγματικά όταν ξεκινήσαμε δεν επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη κάτι τέτοιο, μια αναφορά σε έναν δεοντολογικό κώδικα. Το να είναι όμως αυτό εφικτό και να μπορέσει να λειτουργήσει ήταν κάτι το οποίο πετύχαμε να γίνει. Και το άρθρο 7 μία από τις οριζόντιες αρχές σας τις αποκαλέσω έτσι που μπορέσαμε να εντάξουμε σε διαφορετικά σημεία. Η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της ισότητας των φίλων. προς πελασιμότητα όσον αφορά άτομα με ειδικέ ανάγκε. Ε, ε, σε σχέση με τους διαφορετικού σκιώδη εισηγητές ή εισηγητές των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών μπορούσαμε να σημειώσουμε συνένεση για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό και για το 8 το ίδιο πάλι βιοπικιλότητα, προστασία συστημάτων καταφέραμε να το συμπεριλάβουμε ήταν ένα από τα κυριότερα σημεία που ψηφίστηκε και εντάχθηκε στην εντολή και μετά σε σχέση με τη διαφάνεια, άρθρο 13, πρόσθετη αναφορά σε σχέση με με την ε, πτυχή αυτή όσον αφορά την εντολή μας που ε, μόλις ε, έγινε λόγος λίγο πιο πριν, ένα λεπτό πριν για την έκβαση που πρέπει να επιτυγχάνεται με λιγότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση κατά την επόμενη περίοδο σχεδιασμού. Επόμενο άρθρο, το άρθρο 14 και πάλι εκεί αναγκαστήκαμε να υπαναχωρήσουμε τώρα για το όνομα των πέντε ταμείων, τον, τον, τον τίτλο των πέντε ταμείων που είχαμε συμπεριλάβει. Τώρα εδώ σε σχέση με την ε, Συμφωνία για την Εταιρική Σχέση αναγκαστήκαμε να υπο, υπαναχωρήσουμε. Ο όρος σύμβαση ή συμβόλαιο δεν γινόταν δεκτός. Υπήρχε κόκκινη γραμμή για τα κράτη-μέλη σε αυτό το σημείο. Θεωρούν ότι αυτό δεν βρίσκεται στη φύση των πραγμάτων από πλευράς κρατών και για την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί έτσι να επηρεάσει και να διαμορφώσει τα πράγματα. Κατά τούτο λοιπόν υπήρξε μια τροποποίηση όσον αφορά αυτό το σημείο. Και μετά κάνουμε λόγο και συμφωνήσαμε για την ε, αναγκαία αναθεώρηση όπου αυτό θα απαιτεί το. Επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη σε αυτή την εταιρική, ε, συμφωνία εταιρική σχέσης να υπάρχουν λιγότερα σημεία που θα παριθμούνταν, θα παριθμούνταν. και ευθύ εξ αρχή ε, είπαμε εμεί ότι θα θέλαμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο έγγραφο στο οποίο θα μπορούσαμε εξειδικευμένα να αναφερόμαστε σε εκείνα τα σημεία που θα θέλαμε να ενταχθούν και να συναπαρτίζουν αυτά τα σημεία αυτή τη συμφωνία για την εταιρική σχέση. Ε, δηλαδή ολοκληρωμένη συμφωνία και να δούμε ποια σημεία θα μπορούσαν να εξεταστούν με μεγαλύτερη ελαστικότητα σε μια υστερότερη φάση όταν θα περνούσαμε στα λειτουργικά προγράμματα, στην εφαρμογή τους. Αυτό σε σχέση με το 14, σημαντικό. Μπορέσαμε να επιτύχουμε μια συμφωνία για την νέα δομή, άρθρο 15, πώς να υιοθετηθεί και να εγκριθεί η αναθεώρηση λοιπόν αυτών των συμφωνιών ε, ε, εταιρική σχέση. Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε επί πρακτικών σημείων και η παρασκευή του άρθρου 23 είναι και αυτή σημαντική υπόθεση ε, το, ε, ο προγραμματισμός ε, όσον αφορά την δράση των κονδυλίων αυτών, των ταμείων αυτών σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο διασφαλίστηκε όπως επιθυμούσε η Ευρωβουλή και τώρα σε σχέση με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται προς την, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Και πάλι απόλυτη συμφωνία επ' αυτού. Άρθρο 24, απλά για να το αναφέρω, περιεχόμενο προγραμμάτων αναφέροντας τώρα τη συνεισφορά των προγραμμάτων. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες που θα συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις ε, περιφερειακές στρατηγικές όπου γίνεται λόγος για αυτές τις συμφωνίες ε, όταν είχαμε το θέμα των ορισμών για παράδειγμα. Και πάλι εδώ για τους δείκτες που θα χρησιμοποιούνται μέσω των οποίων θα μπορούμε να καθορίζουμε αυτές τις δράσεις και να τις αξιολογούμε. Μετά ένα άλλο σημείο στο 25 που συνεχίζω με κάποια άρθρα στη συνέχεια τώρα. Το 25 είναι το άρθρο εκείνο για την τον οριζόντιο συμβιβασμό όσον αφορά την προσέγγιση του κοινού στρατηγικού πλαισίου και η, εσείς η κυρία το γνωρίζει αυτό ακριβώς που μπορούν να ε, εγκριθούν αυτά πριν από την έγκριση της εταιρικής σχέσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Στη συνέχεια το άρθρο 26 διατάξεις αυτού του προγράμματος, διαβάζοντας, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκάρσιες, τις οριζόντιες αρχές ε, που ισχύουν στα 5, 7 και 8 άρθρα. Το άρθρο κλειδί τώρα, το 87 σε σχέση με το 87 για τα λειτουργικά προγράμματα. Πρόκειται για το περιεχόμενο έγκριση, προσαρμογή, τροποποίηση κτλ. Και πάλι εδώ το Συμβούλιο ήθελε να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα σε αυτό το άρθρο. Τι πρότειναν. Πρότειναν την ιδέα ενός διαχωρισμού στα λειτουργικά προγράμματα. Μπορέσαμε πολύ εξειδικευμένα να δούμε και να εξετάσουμε υπολογίζοντας το τι θα μπορούσε με διαφορετικό τρόπο να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης σε μια συμφωνία εταιρική σχέσης. Μπορεί κάποια από αυτά να τα διαβάσετε. Το άρθρο 93, τα πιλωτικά προγράμματα για παράδειγμα, που μειώθηκαν από, σε 5 εκατομμύρια από τα αρχικά 10 εκατομμύρια που είχαν προταθεί Ίσως αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για όλο αυτό το πλαίσιο. Ερώτηση τώρα είναι. Κάναμε εμείς όλες αυτές τις συζητήσεις. Είχαμε 12 τριμερείς διαλόγους. Είδαμε πώς λειτουργήσαν τα πράγματα και με όλους αυτούς τους διαλόγους είχαμε παρακολουθηθεί από τους σκιώδεις εισηγητές Τώρα, το ότι καταλήξαμε σε συμβιβασμούς που είναι αποδεκτοί στο τέλος, γι' αυτό είπαμε ναι και δεχθήκαμε. Και δεχθήκαμε την προσέγγιση για τον δεοντολογικό κώδικα που συμπεριλαμβάνεται τώρα σε αυτό το έγγραφο. Και γι' αυτό είχαμε και ένα πρόσθετο κείμενο επιπλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η διάσταση. Συμφώνησε και το Συμβούλιο και είχαν κάποιο άλλο κείμενο από πλευρά τους ε, για την ε, αναδρομική ας το πω έτσι πτυχή επ' αυτών μπορώ πραγματικά να πω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει δεκτό διότι έχουν ξεκινήσει, ξεκινούν τώρα τα κράτη-μέλη να προετοιμάζουν αυτές τις εταιρικέ ε, συμφωνίες από πλευρά τους. Αυτό πρέπει να γίνει, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν όλα αυτά το 2014 και ήθελαν να μην υποστούν κυρώσεις και πληγούν, να μην υποστούν πλήγματα αν σε κάποια τμήματα αυτή της προπαρασκευής όπου υπάρχει κάποια συμφωνία να μην πρέπει να τροποποιηθεί, να αλλοιωθεί, να αλλάξει τελικά γιατί θα υπάρξουν ε, ευαίσθητες ε, χρηματοοικονομικές επιπτώσεις αν γίνει κάτι τέτοιο. Είναι συνετό, λογικό κάτι τέτοιο. Δεν είναι δικό μας κείμενο, δεν το επινοήσαμε εμείς αυτό. Το είπαν τα κράτη-μέλη, το πρότειναν και είπαν εντάξει ας μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προπαρασκευή μας αυτή, δώστε μας αυτή τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με αυτές τις δράσεις, να το εντάξουμε στο έγγραφο. Εντάξει, αυτό έγινε. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα κάνουμε λόγο για ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο με την Ιρλανδική Προεδρία και κάνουμε λόγο για θεματική, θεματολογική επικέντρωση και εξετάζουμε πολύ εξειδικευμένα αυτή την προσέγγιση, ιδιαίτερα όσον αφορά το 4 και το 7 που πρέπει να γίνουν δεκτά υπό το πρίσμα των προτάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμα αυτά. Είχαμε μόνο πρώτε διαβουλεύσει επ' αυτών. Επίση και για το ESF, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και εκεί υπήρξαν εξελίξει, υπήρξαν διαπραγματεύσει που διεξήχθησαν ήδη κατά το παρελθόν, παράδειγμα σε σχέση με την Επιτροπή Απασχόλησης, τα είδαμε όλα αυτά και έχουμε συνειδητοποιήσει κατά το μέγιστο ότι εμείς τουλάχιστον οι εισηγητές ότι στο ευρύτερο αυτό πρίσμα που πρέπει να υιοθετήσουμε. Μπορούμε επί της ουσίας να δεχθούμε αυτά τα οποία είχαν ενταχθεί, είχαν προταθεί σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ένα πράγμα αυτό, ένα πράγμα για τις δαπάνες πράγματι το Συμβούλιο πρότεινε ένα άλλο ποσοστό το οποίο θα πρέπει να ε, στοχεύει και να καλύπτει τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις διάφορες τομεακές κατηγορίες που θα υποστηριχθούν, θα ενισχυθούν. Εμείς από την άλλη πλευρά στο δικό μας κείμενο είχαμε προσεγγίσει μεγαλύτερη ελαστικότητα. Δηλαδή είχαμε πει ενδεικτικά να ισχύει αυτό το χ ποσοστό, για παράδειγμα, σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείναμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κάποιε ιδέε εκείνη από πλευρά τη. Διότι είναι μια πραγματικότητα αυτή η μία πλευρά των δαπανών σε σχέση με τι χώρε μα, τα κράτη-μέλη και ένα νέο ποσοστό που προτείνεται από το Συμβούλιο. Πώ θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση, να υπήρχε μια συνεισφορά ω πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Άντορ να πρότεινε κάτι, του ζήτησα να μπορέσει να υποβάλει μια πρόταση, να δούμε πώ μπορούμε να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον σε σχέση εμεί με την εντολή μα και εκείνο με την πρόταση για το ποσοστό, πώ θα μπορούσε να γίνει. Το είδαμε, το εξετάσαμε άρθρο ανά άρθρο σήμερα και δεν θα χρειαστεί ίσω ενδεχόμενα να επαναληφθεί αυτό το εγχείρημα ε, στο άμεσο μέλλον. Έχουμε το στρατηγικό πλαίσιο, θεματολογική προσέγγιση και όλα αυτά και υπό το πρίσμα όλων αυτών ίσως θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε για την ψήφιση προς έγκριση και να προλιάνουμε το έδαφος με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε. πολύ. Ερωτή σχόλιο Γιάνν Όλμπριχτ. Είχα μια ερώτηση προς τον Λάμπερτ για τον κώδικα δεοντολογίας. Ποιο είναι το επίπεδο συμφωνίας επί του κώδικα δεοντολογίας. Είναι ένα γενικό ερώτημα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πρόεδρος. Άλλα σχόλια, ερωτήσεις. Κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα τα, επειδή μίλησε αγγλικά θα τα πω και εγώ αγγλικά. Λοιπόν, ε, μας είπε πολύ ωραία πράγματα ο συνάδελφος. Ε, φαντάζομαι όμως την ένταση, τη δουλειά, το χρόνο που έχει αφιερώσει. Τον ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά. Ένα σχόλιο, μέσα τον παρατήρηση ουσιαστικά, είναι κάπως ε, οι συνθήκες που έχουμε τώρα και ίσως θα έπρεπε να μας απασχολήσει το κατά πόσον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη Έχω την έκθεσή μου για την πολιτική συντοχή και ενεργειακή πολιτική. Η Ολομέλεια την ενέκρινε στο Στρασβούργο, την τελευταία Ολομέλεια. Είχα στενή συνεργασία με συνάδελφους από την Άλντε και την έκθεση τη στήριξε η ευρύτατη πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Ίσως λοιπόν αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία δέχτηκε το Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Τους πάντων να ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Πρώτος, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος, ο Νίκος Χρυσόγελος και μετά η Κορνέλια Άρνιστα. I haven't understood very well uh, about the... Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπατε για τον κώδικα διοντολογίας και τη συμφωνία, τη συμφωνία εταιρικής Πολύ ε, θα ξέρετε ότι υπάρχει νόμος σε χώρες για τη συμμετοχή των περιφερειών. Δηλαδή για την κατάρτιση των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουμε όμως συζητήσει και κάτι ακόμη εδώ. Η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική. Και υπάρχουν χώρες που δεν την προβλέπουν με νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα των σχεδίων περιφερειακής κατάρτισης. Δεν κατάλαβα πολύ καλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το συμβιβαστικό. Ναι, μεν δεν υπάρχει νομοθεσία ενδεχομένω, αλλά αυτή η διαδικασία συμμετοχής, κοινή συζήτηση, συναπόφαση σε εθνικό επίπεδο με συμμετοχή των περιφερειακών αρχών, περιφερειακών συμβουλίων, κοινωνίε των πολιτών, πριν την τελική κατάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων είναι κάτι που υπάρχει. Πριν συμφωνεί δηλαδή το κράτο μέλο με την Κομισιόν. Ή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη συμφωνία. Ε, Κορνέλια Έρνστ. Η Κορνέλια τετοιο σε συμφωνια Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, μάλλον όλους τους εισηγητές, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Μία ερώτηση έχω. Ο κύριος Φανλιστελρό είπε στο τέλος ότι υπάρχει υποστήριξη, για τα, αλλά δεν μιλήσατε για ποσοστά. Είπατε για τα ποσοστά δεν έχουμε καταλήξει. Τι ακριβώς συζητείτε, στελεστής φτώχειας ή συζητώνται άλλα ποσοστά, υπάρχουν άλλες συζητήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάποιον άλλον συνάδελφο. Οπότε να παρακαλώ τον Λάμπερτ να απαντήσει. Ο κ. Αντλής Τελρό, αρχίζω από το τελευταίο ερώτημα για το ΕΚΤΑ για το Κοινωνικό Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση. Το θέμα είναι ποιο μέρος των κονδυλίων θα αποδοθεί στο ΕΚΤ. Περί αυτού του ποσοστού μιλάμε, είναι το μόνο ποσοστό για το οποίο γίνεται συζήτηση. Και έπειτα έχουμε το Συμβούλιο, το οποίο έχει κάνει μία πρόταση για μία διακύμανση για την εφαρμογή που είναι διαφορετική από την πρόταση της Κομισιόν. Εμείς ως Κοινοβούλιο είπαμε ότι ενδεικτικά ακολουθούμε τα ποσοστά της Κομισιόν. Δηλαδή έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς πρακτικά μπορούμε να το εφαρμόσουμε, αλλά είναι το μόνο ποσοστό το οποίο έχει συζητηθεί. Ουσιαστικά είναι δύο τα ποσοστά που είναι και στο δικό μας, στη δική μας εντολή και στην εντολή του Συμβουλίου. Και όπως είπα και πριν, ελπίζουμε και περιμένουμε ο κύριος Άντορ να μας παρουσιάσει κάποιες ιδέες για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό τα επόμενα χρόνια, αλλά προς το παρόν είμαστε σε διαρευνητική φάση. Διερευνούμε δηλαδή τα ενδεχόμενα και προσπαθούμε να συμφωνήσουμε. Υπό αυτήν την έννοια είμαστε ήδη στη φάση όπου έχουμε συμφωνήσει για το σύστημα για την ε, περίοδο αυτή. Δηλαδή μπορεί κάθε χώρα να προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση αν το συνολικό ποσοστό. Βέβαια έχει το έχει φτάσει σε κάποιο σημείο της περίοδου. Το θέμα είναι τι θα ε, συμφωνήσουν συμβούλοι και Κομισιόν. Εμείς προσεγγίζουμε περισσότερο τη θέση της Κομισιόν και όχι τόσο του Συμβουλίου προς το παρόν. Τώρα, για το άρθρο 5, τι έχουμε συμφωνήσει. Εμείς παίρνουμε την αρχή της εταιρικής σχέσης ε, ως βάση. Και φυσικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Δεν έχει τόσο σημασία πώς είναι οργανωμένη κάθε χώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό. Οι πλεγμένοι φορείς θα πρέπει να τηρήσουν τα στοιχεία τα οποία εμείς τους έχουμε δώσει. Υπάρχει μία σειρά, υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι κανονισμοί που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Είναι πλοκά τα πράγματα βέβαια, αλλά αν θέλουν τα κράτη να πάρουν τα κονδύλια για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, θα πρέπει να επεξεργαστούν αυτά τα προαπαιτούμενα και να τα λάβουν υπόψη τους. That's the answer. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορώ να μπω σε μεγαλύτερο βάθο. Και φυσικά υπάρχει και αρχή τη επικουρικότητα, Γιατί είναι ευθύνη των κρατών μελών Φυσικά επαναλαμβάνω ότι πρέπει να υπάρχει προετοιμασία και προπαρασκευή μαζί με όλους τους άλλους εταίρους. Ερώτημα του κυρίου Όλμπριχτ για τον κώδικα δεοντολογίας. Code of Conduct. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το βασικό σημείο είναι να έχουμε αυτόν τον κώδικα διοντολογίας. Το δεύτερο είναι πώς θα έχουμε έναν κώδικα διοντολογίας. Με τη μορφή μιας κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτή είναι η απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω συμφωνήσαμε, θα προτείνει ένα κείμενο, ή μια κατεξουσιοδότηση πράξη και στο σημείο 5, εδάφιο 3, υπάρχει μια διάταξη όπου προβλέπονται τα βασικά στοιχεία. Το Συμβούλιο δέχεται τον κώδικα διοντολογίας και τη συμφωνία εταιρικής Γι' αυτό σας έδωσα κάποιες πληροφορίες Υπάρχει μια δήλωση που έχει προσθεθεί στο νομικό κείμενο. Αυτό ήταν απαραίτητο για να μην έχουμε αργότερα εκπλήξεις. Το δέχτηκε το Συμβούλιο. Και έχουμε λοιπόν την αναφορά σε αυτή τη δήλωση. Είναι λοιπόν κάτι που γίνεται αποδεκτό από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και αργότερα θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένη κατεξουσιοδότηση πράξη. Η κυρία Κολάρσκα Σκαμπομπίνσκα έφυγε, αλλά τα είπε πάρα πολύ σωστά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια εντολή και αυτό έρχεται πρώτο, η εντολή μας. Και όπως συζητήσαμε και μαζί με τον Μάρκους Πίπερ στη δική του έκθεση για το μέσο διασύνδεση. εάν χρειαστεί αλλάζουμε την εντολή. Αν δηλαδή προκύψει ανάγκη, αλλάζουμε την εντολή, αλλά παρακαλώ ε, πρέπει πρώτα να μου το πείτε. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο τουλάχιστον άμεσα. Απ' την άλλη βέβαια, αν υπάρχει μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία, όπω αυτή τη κυρία Κολάσκα Μπομπίσκα, η οποία έχει εγκριθεί, φυσικά και μπορεί να πειράσει τι συζητήσει μα. Όταν συζητάμε τα επιμέρου άρθρα ή και όταν ψηφίζουμε τελικά αργότερα στην Επιτροπή μας το τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά και υπάρχει πάντοτε δυνατότητα επιρροή, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή η εντολή. Γιατί αυτή είναι η μόνη βάση που έχουμε. Η εντολή μα, επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε να εργαστούμε έτσι, σε αυτή τη βάση. Και επαναλαμβάνω ότι στην όλη διαδικασία μπορείτε να συμμετέχετε. Όλοι. Οι εισηγητές, οι ε, θεωρούν ότι αυτό που έχουμε συμφωνήσει μέχρι στιγμή, μπορεί να είναι αποδεκτό. για τα σημεία των οποίων έχουμε εν μέρη τουλάχιστον συμφωνήσει, δεν νομίζω να κατάλαβα από τους συναδέλφους ότι υπάρχουν ενστάσεις, ότι διαφωνούν. Θα δούμε. Αυτό που είπε η κυρία κολασκα Κολάσκα-Μπομπίνσκα είναι εύκολο να το λέει κανεί. Εντάξει, ήταν πράγματι σκληρέ οι διαπραγματεύσει. Είναι αλήθεια αυτό. Τελικά όμω, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, τότε να ευχαριστήσω τον uh, Λάμπερτ για όλες αυτές τις πληροφορίες και να πω στους συναδέλφους, ιδίως uh, σε όσους δεν έχουν εμπλακεί σε αυτές τις uh, διαπραγματεύσεις, τις διοργανικές, ότι το κείμενο αυτό το οποίο σας έχουμε δώσει είναι ένα κείμενο με τέσσερις στήλες όπως σας είπα και είναι ένα εσωτερικό έγγραφο των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Το έγγραφο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αντικατοπτρίζει τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα. Όσον αφορά το στρατηγικό προγραμματισμό, έχουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη διαπραγματευτική ομάδα ουσιαστικά, καθώς επίσης και από το Συμβούλιο. Πρόκειται όμως να τροποποιηθούν ενδεχομένως μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Ξέρετε ότι α, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να έρθει τελική έγκριση. Αυτό ισχύει λοιπόν και για το εσωτερικό αυτό έγγραφο με τις τέσσερις στήλε και ιδίω για τα όσα λέγονται στην πρώτη στήλη. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα εναπόκειται σε περαιτέρω αλλαγές, ενδεχόμενες αλλαγές. Να το γνωρίζετε αυτό, όταν επεξεργάζετε το κείμενο αυτό ή το χρησιμοποιείτε ή το παρουσιάζετε σε άλλους συναδέλφους σας ή στις δικές σας τις περιφέρειες. Βρίσκεται, είναι ένα κείμενο το οποίο βρίσκεται ακόμα σε μια φάση εξέλιξης και περαιτέρω διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε στη δύσκολη αυτή διαδικασία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχά, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο τη διαδικασία αυτή που κατέληξε τελικά πολύ νωρί σε ένα κείμενο, προσπαθώντα τελικά να καταλήξουμε στα λειτουργικά προγράμματα και συμφωνίε εταιρική σχέση. Προφανώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρέσει και το σε ορισμένα πράγματα περισσότερο, θα ήθελα να δει κάποιε αλλαγέ σε κάποια άλλα, ωστόσο θεωρούμε το κείμενο καλά ισορροπημένο. ευχαριστήσουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί υπεραμήθηκε κάποια σημαντικά στοιχεία της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία ακούσαμε. Μία από τις δεσμεύσεις που έχουμε στην Διοργανική Συμφωνία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσίαζε περισσότερες πληροφορίες για τον κώδικα συμπεριφοράς, τον δεντολογικό κώδικα. Αυτό έγινε. Νομίζω ότι σας δώσαμε τις περισσότερες αυτές πληροφορίες και σε εσά αλλά και στα κράτη-μέλη και τα στοιχεία αυτά τα επιπρόσθετα θα συζητήσουμε πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Όσον αφορά τώρα την συμμετοχή των περιφερειακών αρχών, να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Βανίστερο. Στο άρθρο 5,1 στα πλαίσια της συμφωνίας υπάρχει ένα νέο στοιχείο το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν εταιρική σχέση με τοπικές περιφερειακές αρχές. Αυτό είναι επιπρόσθετο σε σχέση με αυτά που είχε προτείνει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι αποσαφηνίζεται περισσότερο το σημείο αυτό πλέον με την περαιτέρω πληροφορία. Τώρα, όσον αφορά τώρα το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο θεωρούμε βρίσκεται πιο κοντά σε εμά από ότι το Συμβούλιο. Η βασική ιδέα είναι ότι ιδίως στην χρονική αυτή στιγμή των οικονομικών δυσκολιών Χρειαζόμαστε μια πραγματική κριτική μάζα πόρων που να μπορεί να επενδυθεί στους ανθρώπους, στους ανθρώπινους πόρους. Αυτή είναι η βασική ιδέα που βρίσκεται πίσω από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ιδέα αυτή στις περαιτέρω συζητήσεις που θα γίνουν στον τριμερή διάλογο. Και μια τελευταία παρατήρηση αναφερόμενο στην Ιρλανδική Προεδρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Ιρλανδική Προεδρία δεσμεύτηκε να επιτευχθεί μια συμφωνία για το όλο πακέτο πριν το καλοκαίρι. Θα θέλαμε ειλικρινά να υποστηρίξουμε το έργο της δικής σας Επιτροπής και τη δική σας συμβολή προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Άκουσα ότι είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρέσκεται σε κάποια σημεία ενώ κάποια δεν τα βρίσκει τόσο καλά. Αλλά από ό,τι φαίνεται συμφωνείτε με όλα και αυτό είναι πολύ θετικό. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ο Λάμπερτ είπε ότι, είπε ε, ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία, το οποίο θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε ακόμα περισσότερο, δεχομένω να είναι το τελευταίο σημείο που θα επικυρωθεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Μετά το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου θα δούμε αν ε, έχει αλλάξει καθόλου η στάση του Συμβουλίου. Πάντως νομίζω ότι το συγκεκριμένο αυτό σημείο θα είναι αρκετά δύσκολο. Συμφωνώ επίσης με αυτό το οποίο υπόθηκε ότι τις δύσκολες αυτές στιγμές χρειαζόμαστε πραγματικά πολλά κονδύλια τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που υφίστανται σε κάποιες περιφέρειες, ιδίως αυτές οι οποίες περνάνε από, τη, από την κατηγορία της στην πιο πάνω κατηγορία και για τις οποίες ουσιαστικά μειώνεται η χρηματοδότηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές, οι οποίες βλέπουν πολύ σημαντικές μειώσεις, πολλές φορές στις τάξεις του 12-15%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πραγματικά απειλεί και την ίδια τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων, την απορρόφησή τους. Η ευελιξία λοιπόν αποτελεί μια πραγματική πρόκληση, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να επενδύσουμε σε ανθρώπινο κεφάλαιο, απόλυτη αναγκαιότητα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα πρέπει να κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η αποτελεσματικότητα των κονδυλίων αυτών. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να βρούμε το κατάλληλο επίπεδο ευελιξία που θα μα επιτρέψει να είμαστε τελικά αποτελεσματικοί. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό όσον αφορά τον γενικό κανονισμό τη κοινέ διατάξει και μπορεί να ξεκινήσουμε τώρα με την συνεδρία των στονιστών. Παρακαλώ όσοι δεν συμμετέχουν στην συνεδρία των στονιστών να αποχωρήσουν από την αίθουσα. And I hope that all the are here. Και ελπίζω να είναι παρόντες όλοι οι συντονιστές ή τουλάχιστον να είναι καθοδόν. Μπορεί κάποιος παρακαλώ πολύ να καλέσει τον Φρασό Αλφονσί.